Uh, uh, uh, Καλησπέρα, συναδελφοί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Με πρώτο το 51. Απαλλαγή. Και παρουσίαζει ο εισηγητής, τον οποίο δίνω και το λόγο, δηλαδή σε μένα. Τα καλά νέα πρώτα. Ξανά άνοιξε το γυμναστήριο σήμερα του Κοινοβουλίου. Ίσως και γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς συναδέλφους παρόντες. Θέλουν να εξασκηθούν πριν έρθουν στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Επίσης, ξεκινώντας, θέλω μερικές γενικές παρατηρήσεις να διατυπώσω. το θέμα της ευθύνης και της νομιμότητας και η χρηματοδότηση των ε, κονδυλίων της χρηματοδότησης από τις πολιτικές ομάδες που θίξαμε εντάχει σήμερα. Θα διατυπώσουμε γνωμοδότηση. Ωστόσο πριν από αυτό, ασφαλώς θα θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε το θέμα τη οικονομικής διαχείριση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων μας στο Κοινοβούλιο. Επίσης, ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, των ε, ελεγκτών μάλλον, θα δείτε από το σχέδιο έκθεσης, ότι από τις 20, ε, 6 ή 20 ε, δράσεις θεωρούνται μη ίσονος σημασίας, ίσονος κινδύνου. Θα μας πούν λίγο οι εσωτερικοί ελεγκτές τις λεπτομέρειες για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου αναθεώρηση των ε, ποσών αποζημίωσης για τις αποστολές των πιστοποιημένων βοηθών. Σημαντική βελτίωση και έτοιμε βεβαίω ότι θα συμφωνήσουν, θα πούν μάλλον οι ίδιοι ότι θα χρειαστούν περισσότερη, ε, μεγαλύτερη αύξηση. Επίσης το θέμα των ασκουμένων που δεν μπορούν να λάβουν προκαταβολή στα έξοδα των αποστολών. Είναι ένα σημαντικό θέμα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προκαταβολή ε, αυτών των εξόδων για τους ασκουμένους, ώστε να μην χρειάζεται οι ίδιοι να προκαταβάλουν τα ποσά, το έχω επισημάνει και στην έκθεσή μου. Στα επιμέρους, θα είδατε στο σχέδιο εκθέσης αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εξετάζω χωριστά τις γενικές ευθύνσεις με σχόλια για την καθεμία παραδείγματι. Εδώ επισημαίνω την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που σημειώνει πως υπάρχει μια αύξηση στις θετικές εντυπώσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευπρόσδεκτο, προσωπικό Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι προάγεται πάντα ε, το θέμα των ίσων ευκαιριών στη διαχείριση, στην πολιτική διαχείριση των ανθρωπινών πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δε τις περιπτώσεις ε, παρενόχλησης. Πολύ σημαντικό αλλά και επίκαιρο πρόσφατα, ευπρόσδεκτη η πρόταση του Γενικού Γραμματέα για την εισαγωγή ενός δικτύου απόρριτης παροχής συμβουλών από συμβούλους στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ε, είτε βοηθός, είτε ασκούμενος, είτε οποιοδήποτε εργάζεται σε βουλευτές ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού. Υποδομές και επιμελητεία. Μιλώ ιδιαίτερα για το θέμα της πολιτικής για τα κτίρια. Μια στρατηγική για τα κτίρια λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία ωστόσο αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολο σε χρονιά Brexit να καλυφθεί το θέμα αυτό. Βέβαια υπάρχουν και όλα τα θέματα τα σχετικά με τα της του PHS, του Polar Pack. Είναι θέματα που συστήνει ακόμα το Προεδρείο, πρέπει να καταλήξουν σε μια επιλογή που θα είναι είτε να μην αναλυφθεί δράση, είτε να, ανακαινιστεί, ε, είτε να ανοικοδομηθεί το κτίριο και μέχρι ότου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις θα είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για μια συνολική στρατηγική για τα κτίρια. Πάντως είναι σημαντικό κάποια στιγμή να έχουμε μια γενική στρατηγική για τα κτίρια, να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και ποια είναι τα κτίρια που έχουμε διαθέσει μας στο μέλλον. Επίσης, διερμηνία και διασκέψεις, όπου σημειώνω πως ο συνολικός χρόνος διερμηνίας στις υπηρεσίες διερμηνίας για τους διερμηνείς από τις 11,54 ώρες έχει αυξηθεί στις 13,25 και αυτό που έχω να πω εδώ είναι ότι η αδίποτε αλλαγή στις συνθήκες εργασίας θα πρέπει να προκύψει κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των συνδικαλιστικών ενώσεων και του Γενικού Γραμματέα και βεβαίω θα μεριμνήσουμε σε αυτή η συνεργασία και στο μέλλον να συνεχιστεί εφόσον πρόκειται να προταθούν νέες αλλαγές. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, η Σύμβαση για την υπηρεσία, για τις υπηρεσίες ταξιδίων εκπνέει και προεκπεί να ετοιμαστεί η προσεχή, εκπνέει στο τέλος του 2018, ετοιμάζεται ανοιχτή προσγλώση υποβολής προσφορών για την επιλογή του νεοδιοξιδοτικού γραφείου. Ιδίως μας ενδιαφέρει η τιμολόγηση, γιατί είχαμε στο παρελθόν διάφορα σχόλια ότι ήταν πολύ πιο υψηλές οι τιμές που πρότεινε το ταξιδιωτικό γραφείο από κάτι που θα μπορούσε να βρει κανείς είτε στο διαδίκτυο είτε σε ένα άλλο πρακτορείο. Επίσης σημειώνω ότι θα πρέπει στην προσεχή σύμβαση να προσφέρονται διαθέσιμες υπηρεσίες και κατά το Σαββατοκύριακο, γιατί σε Σαββατοκύριακο είναι πολύ δύσκολο και δικυριακή να αλλάξει κανείς το εισιτήριό του ή να ζητήσει ένα εισιτήριο. Το έχω προσωπικώς αντιμετωπίσει αυτό και στη νέα σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται κάτι σχετικό με την διαρκή διαθεσιμότητα του κέντρου κλήσεων τη ακτική υπηρεσία ακόμη και τα Σαββατοκύριακα για κρατήσει ή αλλαγέ. Σχόλια έχω περιλάβει επίση για τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομία και Τεχνολογική Υποστήριξη, όπω επίση και για τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλεια και Προστασία. Θα δουν οι συνάδελφοι τα σχόλιά μου στο σχέδιο τη έκθεση που σα έχει διανεμηθεί. Σχόλια έχω επίση για την εξασφάλιση ενό φιλοπεριβαλλοντικού κοινοβουλίου με ικανοποίηση σημειώνουμε πως το Προεδρείο έθεσε εφαρμογή το σχέδιο για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ένα σχέδιο για μετάβαση σε ηλεκτρικό στόλο αυτοκινήτων. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο εγγύς δυνατόν μέλλον να εξασφαλιστεί αυτό. Ε, επίσης, ένα-δύο πράγματα που δεν έχω αναφέρει στην έκθεσή μου και θέλω προφορικά να τα σχολιάσω είναι γενικές δαπάνες, αποζημίωση γενικών δαπανών, την οποία δεν ε, θίγω προς το παρόν, καθώς γνωρίζουμε ότι μια ομάδα εργασίας μεικτή από όλες τις ομάδες ε, εξετάζει το θέμα αυτό και περιμένουμε τις συστάσεις της κάπου το Μάρτιο. Πρόταση που ελπίζουμε ότι θα έχουμε πριν να καταλήξουμε στις δικές μας τροπολογίες, εάν δεν έχει όμως υποβληθεί μέχρι τότε. Ασφαλώς θα περιληφθεί στο κείμενό μου παράγραφος ε, για το θέμα της αποζημίωσης γενικών εξόδων που ξέρουμε ότι έχουν, ε, έχει απασχολήσει τους αδέρφους και στην απαλλαγή στο παρελθόν επανελειμμένος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το παραλείψουμε. Αλλά είναι σημαντικό θεωρώ. Πρώτα να δούμε τις προτάσεις και μετά να κάνουμε σχόλια. Ένα άλλο θέμα που δεν έχω θίξει, αλλά ίσως να σας ενδιαφέρει, Μπάρτ είναι το σύστημα της εκούσιας τάξης. Δεν το φύγω γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Γενικός Γραμματέας πρόκειται να διατυπώσει προτάσεις σύντομα για το θέμα αυτό. Και ίσως θα πρέπει να έχουμε τις προτάσεις πρώτα. Ελπίζω να τις έχουμε πριν να καταλήξουμε στο σχέδιο. Αν όχι, θα συμπεριλάβω μια παράγραφο, ένα κείμενο σχετικό με το τμήμα αυτό. Αλλά πρώτα ήθελα να, ακούσω τα, να διαβάσω τα σχόλια και τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα. Όπως είπα, εάν δεν γίνει ανακοίνωση εγκαίρως, τότε θα περιλάβω εγώ τα δικά μου σχόλια στο κείμενο της έκθεσης. Αυτά από μένα και την έκθεσή μου. Κύριε Πρόεδρε, που είμαι εγώ ο Πρόεδρος, και βεβαίως περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων και τη συζήτηση με τους κοιόδης για να διευθετήσω οποιαδήποτε επιφύλαξη μπορεί να έχουν. Αυτά για την έκθεσή μου και προχωρώ αμέσως στους σκιώδεις και δει την κυρία Σμιτ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη αυτή η έκθεση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να οικοδομήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα ε, καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες. Ε, να είναι σύντομη Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κάθεστο των Βρετανών υπαλλήλων γιατί νομίζω ότι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση και λογικό είναι να θέλουν κάποια διασφάλιση αλλά ρεαλιστικά πρέπει να δούμε το τι θα διαπραγματευτεί η Κομισιόν με τις ε, κυβερνήσεις. Επίσης, όπως είπατε, η DigiCom ε, προετοιμάζει την νέα ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να είναι πιο φιλική προς τον χρήστη και επίσης ε, και τα κοινωνικά μέσα και Πρέπει επιγόντω να δώσουμε περισσότερο βάρο εκεί. Η Γενική Διευθυνσία ΙΤΕΚ e εξακολουθεί να έχει προβλήματα και σε και σε κάποια τμήματα κτηρίων στο Στασβούργο και θα πρέπει να λειτουργήσουν το σύντομο το δυνατόν. Το MEP Portal επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο, βρίσκουμε πληροφορίες Ταυτόχρονα έχουμε την εντύπωση πως υπάρχει μία μεταβάση των δραστηριοτήτων στους βουλευτές και τα γραφεία. Δηλαδή καλή απλοποίηση για την διοίκηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να μεταβάζεται αλλού η δουλειά. Δεύτερον, θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση στην οποία έχουμε βλάβει στα δίκτυα του Κοινοβουλίου όπως είχαμε προσφάτως. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι γίνεται ακριβώς για να υπάρχει αυτή η προστασία ή ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει μια διασφάλιση γιατί υπάρχουν και κόστη όταν πέφτει το δίκτυο. Η Γενική Διεύθυνση SAFE, νομίζω εκπροσωπείται επαρκώς από τα συνδικάτα, έχει μεγάλη σημασία οπωσδήποτε και η προσωπική ζωή των εργαζομένων, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται και η ασφάλεια του Κοινοβουλίου, νύχτες και Σαββατοκύριακα. Μετά τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά, ε, το, τα θέματα των, του Γραφείου Ταξιδίων έχουν ανέβει και οι τιμές και το επίπεδο της εξυπηρέτησης ε, δεν ε, είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά για τους βουλευτές. Μετά ε, αναφέρθηκαν ήδη οι διερμηνείς. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει επίσης είναι τα γραφεία πληροφόρησης τα κράτη-μέλη και εκεί πέρα θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα των, της ισορροπίας των φύλων στην διοίκηση, στις ε, διευθυντικές θέσεις. Ε, υπάρχουν, θέσεις, υπάρχουν γυναίκες ε, που θα πρέπει να καταλαμβάνουν τις θέσεις, όχι επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή έχουν τα προσόντα και μετά έχουμε και το καθεστώς των βοηθών. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ και τον εισηγητή, ο οποίος είναι πάντα στην διάθεσή μας για συζητήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την ε, δομημένη και ισορροπημένη έκθεσή σας για τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016. Η έκθεση αυτή απαντά στο θέμα των βελτιώσεων στην ε, ποιότητα και διαφάνεια των δημοσίων οικονομικών αλλά και στο θέμα της λόγοδοσίας της πολιτικής ηγεσία στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ε, τελικές ε, δαπάνες ε, του 2016 ήταν γύρω στο 19% του τίτλου 5 του ΠΔΠ και γύρω στο 95% από αυτές δεσμεύτηκαν. Ε, βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να απαντήσουμε το πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι πόροι και τι αποτελέσματα επιτύχαμε. Όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2016, την και την κανονικότητα των συναλλαγών θα πρέπει νομίζω να μας ικανοποιεί η άποψη του Ελεκτικού συνεδρίου ότι δεν υπάρχει υψηλότερο επίπεδο σφάλματος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρόταση διορισμού ενός συντονιστή εσωτερικού ελέγχου σε κάθε γενική διεύθυνση δεν θα οδηγήσει σε αυξημένη γραφειοκρατία και φόρτο εργασίας από την πλευρά της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Βλέπουμε πως ε, η Διοργανική Συμφωνία για τη συνεργασία σε ζητήματα προϋπολογισμού και δημοσιονομική πειθαρχία εξελίσσεται ομαλά. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, πληροφορίες για τα συμβόλαια τα οποία δίνονται και για τον τύπο των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως επίσης και για, τις, ε, για τους προϋπολογισμούς των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που είστε και εισηγητής. Ευχαριστώ ε, και για τη συζήτηση που είχαμε ήδη στο Στρασβούργο με τους ε, σκιώδεις. Διάβασα την έκθεση με μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πάντως μια συνεκτικότητα μεγαλύτερη ανάμεσα ε, στην έκθεση αυτή και τις, ε, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Ε, συγκρινόμενο με την προηγούμενη χρονιά που ήμουν εισηγητής, βλέπω ότι υπάρχουν λίγο κάποια επιπλέον ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε και ένα follow-up, μια συνέχεια στα θέματα γιατί βλέπουμε ότι το Προεδρείο κάνει, ε, συνεχίζει, δίνει συνέχεια στα θέματα τα οποία ε, πραγματεύονται τα ψηφίσματα. Το... Ε, τι σημαίνει, σημαίνει ότι το Προεδρείο έχει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερες από ότι η Ολομέλεια έχουν δοθεί, έχουν δοθεί κάποιες... Έχουν παραχωρηθεί κάποιες εξουσίες από την Ολομέλεια στο Προεδρείο, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να αποφασίσουν τα μεμονωμένα μέλη του Προεδρείου εάν και κατά πόσο θέλουν να δώσουν συνέχεια σε κάποια θέματα. Αυτό είναι ε, ε πολιτικό ζήτημα και πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και βεβαίω μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα ε, στα οποία δεν δόθηκα μία συνέχεια. Και πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι ώρες ε, που δαπανούμε εδώ σε αυτήν την ε, Επιτροπή αλλά και το χρόνο που δαπανά η Ολομέλεια για να συζητήσει τα θέματα αυτά <laughs> δεν μπορεί να πάνε χαμένα. Ένα παράδειγμα για να σας δώσω μια γενική ιδέα. Εγκρίναμε α πούμε πριν από λίγο καιρό αλλά και άλλε φορέ όχι μόνο πέρσι, την ιδέα ότι στην προσωπική ιστοσελίδα των ε, Ευρωβουλευτών και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ε, ε, θα υπάρχει μία σελίδα για τους για τους Ευρωβουλευτές και βρίσκει κανείς μία σελίδα με τη φωτογραφία του καθενός μας και θεμητά ο κάθε πολίτης πιστεύει ότι αυτή είναι η ιστοσελίδα μας, αλλά δεν είναι τουλάχιστον μπορούμε να βάλουμε εκεί, σε αυτήν τη σελίδα, οι συνεδριάσεις, να βάλουμε τις συναντήσεις μας, ε, αν έχουμε συναντήσει με του λομπίστε κτλ. Ε, αυτό το είχαμε συμφωνήσει, είχαμε πει ότι θα γίνει σε εθελούσια βάση, οποίο θέλει το βάζει, οποίο δεν θέλει δεν το βάζει, η Κομισιόν το κάνει έτσι κι αλλιώ. Αλλά δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην ε, Χάιτεκ, Γενική Διεύθυνση Χάιτεκ, που μας είπαν, Σα το λέω για λόγους αδιαφάνειας, ε, είπαν ότι μπορείτε να το τροποποιήσετε αυτό το κομμάτι που μιλάει για σας και αν θέλετε το ημερολόγιό σας, δεν ξέρουμε ακριβώς όμως πώς θα το κάνουμε, γιατί είναι ε, περίπλοκο. Και αυτό πρώτη φορά το ακούγαμε και ήταν αντίθετο από αυτά που είχαμε ακούσει μέχρι τότε. Και το δεύτερο είναι Μα είπαν μερικοί, α, η Ολομέλεια θέλει πότε το ένα, πότε το άλλο και συνέχεια αλλαγέ ε, και δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα αυτά για την Ολομέλεια. Μα αυτό είναι όμω σοβαρό και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτή την έκθεση, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια πολιτική φύσεω προβλήματα με τη διοίκησή μα. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε διαρκώ τα μάτια σε αυτέ τι καταστάσει και κάτι άλλο. Έχουμε την ε, ε, δυνατότητα ε, ε, κινδύνου όσον αφορά την φήμη μας. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε θέματα τα οποία συζητήσαμε λίγο πιο πριν σήμερα με τους συντονιστές. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και είναι σαφή. Επομένως, μίλησα και πέρσι στο ελεγκτικό συνέδριο αλλά και στην εσωτερική μας διοίκηση όλοι όλοι ε, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει μία τάση ε, ε, μικρής δειγματοληψίας όσον αφορά τον έλεγχο των ε, δαπανών. Αλλά ο κίνδυνος ε, όσον αφορά τη φήμη μας, που μπορεί να είναι εντονότατος, ιδίω την επόμενη χρονιά που είναι χρονιά εκλογών, ο κίνδυνος αυτός, λέω, είναι ιδιαίτερα μεγάλος και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες συστάσεις και ε, στο ε, ελεγκτικό συνέδριο. Όλα αυτά είναι περίπλοκα και ούτως ή άλλως ε, δεν μπορούμε να ελέγχουμε μόνοι μας τα αριθμητικά στοιχεία και να ψάχνουμε να βρούμε αυτό το ένα λάθος που κάποιος άλλος το παράβλεψε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλω. στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο υπάρχει ε, η δυνατότητα να μελετώνται τα στοιχεία ε, και να βρίσκονται τα λάθη και επομένως ε, θα μπορούσαμε και να το έχουμε και εμείς εδώ. Θα ήθελα να το βάλετε αυτό στην έκθεση. Και επίσης υπάρχουν πολλά μεμονωμένα, όπως ας πούμε το Εθελοντικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο ναι, υπάρχει ομάδα εργασίας, θα δούμε τι θα ε, προτείνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται ή ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τη σύσταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να πιέσουμε τους πάντε μεταξύ άλλων και την ομάδα εργασίας. Επίσης, προβλήματα επικοινωνίας, τα οποία τα αναφέραμε πέρσι ε, και ε, τα, πρέπει να τα αναφέρουμε και φέτος. Ε, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πληροφόρηση, έχουμε προβλήματα όσον αφορά το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα γραφεία της υπηρεσίας πληροφόρησης, πρέπει να είναι το πιο ακριβό σημείο στο Παρίσι, ας πούμε. Ε, πολλά ζητήματα. Θα υποβληθούν βεβαίως κάποιες ε, τροπολογίε έστω και αν ε, όλο το τεχνικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλό, είναι εξαιρετικό, αλλά το πολιτικό κομμάτι χρειάζεται κάποια αρετουσαρίσματα. Ευχαριστώ. Ο Μπάρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντέρικ. Αντικαθιστώ εδώ τον Μπεντικτέ Γιάβορ, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής, αλλά αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται σε τριμερή διάλογο για την οδηγία ενεργειακής ε, αποτελεσματικότητας. Οπότε μου έχει δώσει κάποια πράγματα να πω και θα πω και κάποια δικά μου. Ο Μπένεντικ ε, χαίρεται για το ότι στην έκθεσή σας αφιερώνεται μεγάλο κομμάτι στο Brexit ε, και Αποδέτε μεγάλη προσοχή και εδώ πέρα συμφωνούμε επίσης με αυτό το οποίο είπε ε, και ο Ντένις ότι έχετε γράψει τεχνικά μια πολύ καλή έκθεση αλλά η πολιτική πτυχή θα μπορούσε να ενισχυθεί. Το αναφέρατε και εσείς ε, θελοντικά, συνταξιωτικά ταμεία, αυτά τα οποία κάνει ο Γενικός ε, Γραμματέας. Επίσης υπάρχει αυτό το οποίο λέει ο Μπένεντικ είναι το ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων ήταν αντικείμενο έκθεσης περσινής ε, και εγκρίθηκε πέρσι και ευτυχώς εντωμεταξύ το Πρόεδριο συνέστησε μια ομάδα εργασίας και οπωσδήποτε εμείς ως πράσινοι μαζί με την ΓΚΟΕ θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για το θέμα για να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει μέγιστη διαφάνεια για την αποζημίωση γενικών εξόδων. Δεύτερον, ο Μπένεντικ ε, διαπίστωσε ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει δικαίωμα των βουλευτών να ζητήσουν αποζημίωση για την χρήση αυτοκινήτων στη χώρα τους αυτό προκύπτει από το καθεστώς των ε, βουλευτών, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου έλεγχος. Ε, θα υπάρξει λοιπόν και εδώ σχετική τροπολογία τρίτων. Ο Μπένεντικ θα ήθελε να καταγραφεί ότι θα πρέπει να, υπάρχουν περισσότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ του σταθμού εδώ πέρα Βρυξέλλες ε, Πλάς Λουξεμβούργ και του αεροδρομίου γιατί νομίζω είναι δύο δρομολόγια την ώρα τώρα και να δούμε αν μπορούν να αυξηθούν. Τέταρτον, ο Μπενεντίκ θα υποβάλει τροπολογίες ε, για να περάσει το Κοινοβούλιο σε ε, λογισμικό open source ανοιχτού κώδικα Κατόπιν ε, μπορούν να ενισχυθούν οι παράγραφοι περί σεξουαλικής παρενόχλησης και εδώ πέρα θα υποβάλουμε τροπολογίες. Κατόπιν ο Μπένεντικ ε, θέλει να υποβάλει μια τροπολογία για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ε, για το θέμα των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται τώρα σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έβδομον, Εν τω μεταξύ βέβαια έχει κρυθεί από το Προεδρείο, θα πρέπει δηλαδή να καταργηθούν τα μπουκάλια νερό και να βάλουμε απ' έξω ψύκτες για να μειώσουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Όχι μόνο τους ψύκτες εδώ έξω, αλλά ίσως και εκεί όπου μαζεύονται οι βουλευτές και οι συνεργάτες στα γραφεία τους. 8 η ασφάλεια στο Στρασβούργο του κτηρίου. Ξερίζουμε όταν μπαίνουμε στο ότι υπάρχουν διάφορα κινητά περίπτερα. Αυτό είναι βεβαίως προσωρινή λύση. Θα πρέπει να αναζητηθεί μια πιο κόμψη ε, λύση και οπωσδήποτε θα υποβάλουμε εδώ πέρα τροπολογίες. μετά για αυτό το οποίο είπε και ο Ντένις, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και στις σελίδες των βουλευτών να φροντίσουμε αυτό το οποίο είχε αποφασίσει η Ολομέλεια, δηλαδή να δηλώνονται οι επαφές με τα λόμπια, αλλά και το νομοθετικό αποτύπωμα. Να λέει δηλαδή ο εισηγητής, εγώ συνάντησα τον Χ, τον Ψ και τον Ωμέγα, και είμαι υπεύθυνο για αυτές τις εκθέσεις ως εισηγητής, και εισηγητής κτλ. Και δέκατον, για τους ε, βοηθούς, ο Μπένεντικτ ε, θα υποβάλει τροπολογίες για το δικαίωμα των ε, βοηθών να γίνουν πληροφοριοδότες και κατόπιν ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είναι η αποζημίωση που λαμβάνουν για το Στρασβούργο, η οποία τώρα ρυθμίζεται καλύτερα, αλλά για κάποιους από αυτούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματός τους και αυτό θέλει να το διορθώσει μέσω μιας τροπολογίας ο Μπένεντικτ για να κάνει κάτι ο Γενικός Γραμματέας. Αυτά είναι τα 10 σημεία του Μπένεντικτ. Έχω και τρία δικά μου. Το πρώτο αφορά επίσης τους βοηθούς ήμουν σε μια ακρόαση με τον Κλάου Βέλε. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι από το 2009 και θα συμπληρώσουν δεκαετία, κάτι το οποίο θα επηρεάσει τα συνταξιοδοτικά τους ε, δικαιώματα. Είπε ο Κλάσουελε, δεν μπορώ να κάνω κάτι στην περίπτωση στην οποία δεν έχουν κλείσει κάποιοι δεκαετία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Μετά το αναφέρατε το εθελοντικό συνταξιοδοτικό τομείο, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο Γενικός γραμματέας και με το αν θα φέρει το Μάρτιο προτάσεις, εμείς θα υποβάλουμε σχετικές ε, τροπολογίες. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τα ΜΜΕ. Υπάρχει ένα αναλογιστικό έλλειμμα 370 εκατομμυρίων ε, ευρώ και θα προσθεθούν και άλλοι οπωσδήποτε δικαιούχοι Εν τω μεταξύ ένας ε, δημοσιογράφος του e-Observer έγραψε ένα tweet ότι ρώτησε στην συνέντευξη τύπου της Κομισιόν το τι γίνεται με τη συμμετοχή των ε, Ευρωπαίων ε, Επιτρόπων στο ταμείο αυτό, γιατί δύο από αυτούς ήταν, σύνταξ, ήταν ευρωβουλευτές. Ε, η μία ήταν η Μαριάν Τάισεν, 62 ε, ετών, και ο άλλος είναι ο κύριος Κανιέτε, ο Ισπανός Επιτροπός, ο οποίος είναι 68 ετών ε, και στην ενημέρωση του τύπου φάνηκε ότι ο κύριος Κανιέτε αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά γιατί είχε πληρώσει βεβαίως τις εισφορές του όταν ήταν ευρωβουλευτής και τώρα λαμβάνει κάποια σύνταξη. Είναι αδιανόητο δηλαδή. Πρόκειται για ένα εθελοντικό ε, ταμείο σύνταξης και δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος σύνταξη τη στιγμή που δουλεύει και ως Ευρωπαίος Επίτροπος μάλιστα. Δηλαδή το θέμα δεν αφορά τον ίδιον τον Κανιέτα, ίσως είναι και άλλοι συνάδελφοι που λαμβάνουν ε, λεφτά, ότι είναι πάνω από 63 ετών ε, και λαμβάνουν λεφτά και εργάζονται. Όχι, ε, σύνταξη όταν είναι κάποιο συνταξιούχος και δεν δουλεύει πια, δεν γίνεται αλλιώ. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και είναι και θέμα εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία πρέπει κάτι να κάνουμε και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες. Τέλος, κάτι το οποίο επίσης ε, θα μας απασχολήσει και το είχαμε πει πέρσι, το είχε καλύψει ο Ντένις στην έκθεσή του, το πρόβλημα που υπάρχει δηλαδή με την κατάχρηση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά ιδρύματα, το Προεδρείο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ξεκίνησε κάποιες, ε, να κάνει κάποιες ενέργειες. υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια Πρέπει, δεν ξέρουμε λοιπόν το τι έχει γίνει ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και εδώ πέρα θα υποβάλω τροπολογίες. Αυτά τα 13 σημεία από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ε, I can't see ε. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει το λόγο. Όχι. Ωραία. Ο Μπάρτ κάλυψε τα πάντα νομίζω. Ε, Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο εισηγητή όσον αφορά την ε, ε, την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω σε σχέση με πέρσι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες βελτίωσης ε, όσον αφορά ε, την ε, χρήση των κονδυλίων που έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ανησυχία, προβληματισμό σχετικά με τις διευκολύνσεις ε, που δίνονται και παρέχονται στους ευρωβουλευτές ε, εν ώψη του Στρασβούργου και στα πλαίσια του Στρασβούργου. Δεν ξέρω αν εφήγει ήδη και ζητώ συγγνώμη αν επαναλαμβάνω κάτι. Πιστεύω ότι η Γενική Γραμματεία ε, του Κοινοβουλίου όταν θα έρθει σε διαπραγμάτευση με το Στρασβούργο θα πρέπει να αναφερθεί στην βελτίωση των, της πρόσβασης στο ε, αεροδρόμιο ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό και ότι οικονομικά ε, μπορεί να σημαίνει κάτι τόσο τρομερό, επιπλέον αστυνομική ή επιπλέον σκάνερς. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι μάλλον εύκολο να κινητοποιηθούν κάποια, κάποιες επιπλέον δυνάμεις, κάποια επιπλέον κάποια επιπλέον πόρη. Επίσης, να πω ότι συμμερίζομαι ε, με τα περισσότερα από τα στοιχεία που παρουσίασε ο εισηγητής. Ε, απλώς ε, μία απόχρωση κατά κάποιο τρόπο να δώσω, με ένα μετριασμό. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς με τη σύνταξή του ο κύριος Αρίας Κανιέτε. Δεν ξέρω εάν παίρνει τα χρήματα αυτά, αυτή τη σύνταξη ή όχι. Κατανοώ όμως απολύτως το επιχείρημα γιατί ως ένας ε, ε, επίτροπος έχει πολύ ικανοποιητική ε, αμοιβή, πολύ, πολύ ικανοποιητικό μισθό. Τώρα είναι προσωπική του άποψη, εάν και εφόσον υπάρχει νομικά η δυνατότητα και είναι κάτι νόμιμο να παίρνει τα χρήματα αυτό. Το ζήτημα είναι ε, να ε, ε, καθοριστούν για αυτό το ταμείο συγκεκριμένοι κανόνες. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι κανόνες και δεν αποκλείεται να λαμβάνει κανείς αυτή τη σύνταξη έστω και αν εξακολουθεί να εργάζεται. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Βλέπω κάποια σημεία που νομίζω χρειάζεται να συζητήσουμε, ας κλείσουμε έτσι τη συζήτηση. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Δεν είμαστε τόσο πολύ άριθμοι, αλλά έχουμε πολλά θέματα που εγείρουν οι συνάδελφοι. Και τίνω να συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν στο σύνολό του, κυρίω στα πρώτα σχόλια τη κυρία Σμιτ για το πόσο σημαντικό είναι να μεριμνήσουμε για του Βρετανού υπαλλήλου. Ξέρω ότι του έχουν δοθεί κάποιε διαβεβαιώσει, αλλά πρέπει να το παρακολουθήσουμε. και στη συνέχεια. Σωστά μιλάτε για το νέο ιστότοπο. Θα πρέπει ίσως να ζητήσουμε μια τροπολογία, μια επαλήθευση, μια βελτίωση. Είναι κάπως καλύτερο σχέση με τον παλαιό. Δεν θα ήταν κακό να το κοιτάξουμε και πάλι. Επίσης ε, για την e και τις άλλες γενικές διευθύνσεις και θέματα που προέκυψαν πέρσι όταν ε, κατέρευσε το σύστημα για μια εβδομάδα περίπου. Επίσης, ε, Ρώτημα είναι αν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για το τι θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίζεται ως υπηρεσία προσφερόμενη και ως σύστημα IT. Ποια είναι τα πιο σημαντικά δηλαδή για μας. Να ορίσουμε προτεραιότητες και να καλύπτονται πρωταρχικά τα πιο σημαντικά και μετά τα υπόλοιπα. Για τον κύριο Ντεϊόγκ συμφωνώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε κάποια ενημέρωση για το τι μοίρα είχαν οι συστάσεις. Θέματα επίσης ε, του κυρίου Γιάβα για, την, ε, ε, για τα ταξίδια, για την ασφάλεια, για τους καταγγέλλονται. Ο κύριο Γιάβα φαντάζομαι ότι θα έρθει να καταθέσει, θα, θα, θα προβεί σε καταθέσει τροπολογιών. Τα δύο θέματα του Μπάρτ και του κύριου Ντε θα μας απασχολήσουν λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι για το εκούσιο σύστημα συνταξιδότησης έχουμε δει τα στοιχεία όλοι. Θα θέλουμε να τα κοιτάξουμε όλοι λίγο πιο λεπτομερώς. Βέβαια πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε Ίσως θα είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή να περιμένουμε, να δούμε τι προτάσεις ε, θα καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας, καθώς μας διαβεβαίωνε ότι θα καταθέσει σύντομα προτάσεις. Ας δούμε λοιπόν πρώτα ποιες προτάσεις κατατίθενται και ας σχολιάσουμε μετά. Ιδάλλως, αν δούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και εγώ σκοπεύω να κάνω κάποιες ε, τροπολογίες μέσα από το κείμενο. Για την ε, γενική αποζημίωση και υπόθηκε αυτό και ο Ντένις και εγώ το έχουμε συζητήσει. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαφάνεια. Εμείς οι Βρετανοί μάλιστα δημοσιεύουμε στο μέγιστο δυνατό τις λεπτομέρειες των σχετικών εξόδων, γιατί έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα της ασφάλειας, άλλοι ίσως όχι τόσο, αλλά παντός υπάρχει μια διακομματική ομάδα η οποία πρόκειται να καταθέσει ε, προτάσεις και όταν τις δούμε ας διατυπώσουμε τις προτάσεις μας. Ίσως να μην έχουμε όμως εγκαίρως τις προτάσεις αυτές. Γι' αυτό ήδη εγώ έχω αρχίσει να αναλογίζουμε τι θέματα θέλω να περιλάβω στην έκθεση, όπως σε παραδείγμα συγκεκριμένου κανόνες για τη λογοδοσία, για τις ε, ε, δαπάνες και κάτι άλλο που ασφαλώς θα ενδιαφέρουν τους συναδέλφους και που θα μπορούσαν να τα δεχθούν όλοι. Ε, παραδείγματι ότι δεν πρέπει να μπαίνει σε χωριστό λογαριασμό και ότι θα πρέπει οι βουλευτές να διατηρούν όλες τις αποδείξεις τις σχετικές με τη γενική αποζημίωση και να γίνεται μια εκαθάριση των εξόδων μέχρι το τέλος της θητείας για τον κάθε βουλευτή. Νομίζω ότι είναι θέματα στα οποία μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Ας δούμε όμως η ομάδα εργασία τι πρόταση διατυπώσει. Και αναλόγως να κρίνουμε. Βεβαίως αν θεωρούν συνάδελφοι ότι δεν είναι επαρκεί σε αυτές τι προτάσεις ομάδας εργασίας, θα έχουμε το χρόνο να καταθέσουμε τι τροπολογίε μα. Αυτή είναι η λόγια για τους δεν ε, κατέθεσα σχετικό κείμενο. Αλλά είναι έτοιμο το κείμενο τη δική μου πρόταση. εάν τυχόν και δεν δούμε εγκαίρω προτάσει. Ολοκληρώνω εδώ, σημειώνοντας ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση είναι η 1η Μαρτίου. Περιμένω τους συναδέλφους, περιμένω τις τροπολογίες τους και βεβαίως εάν χρειαστεί κάνουμε τις σχετικές τροποποίησεις. Ευχαριστώ πολύ. Και προχωρώ στο επόμενο θέμα. Απαλλαγή 2016 για τα λοιπά θεσμικά όργανα με τον κύριο Βάλη. Εισηγητή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ντέρεκ. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές, καθώς επίσης και τις γενικές, τους γενικούς γραμματείς των αντιστοίχων θεσμικών οργάνων για τη βοήθεια που έχουν παράσχει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των διοικητικών δαπανών είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά αλλά και για τους πολίτες ε, ειδικότερα. Ε, θα πρέπει με τρόπο αποτελεσματικό να ελέγχεται ε, η όποια δαπάνη χρημάτων ε, και να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τους πολίτες. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω όπως επανειλημμένα υπενθύμηση άλλωστε και ο Στέλφος Μπάρτα αλλά και η πρόεδρος της Επιτροπής ε, και άλλοι που ασχολούνται με το θέμα να υπενθυμίσω λέω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο άμεσα εκλέγεται από τους πολίτες και επομένως ε, ζητά διευκρινήσεις από το Συμβούλιο όσον αφορά τη φύση των δαπανών του και με αυτή την έννοια είναι σαν να υποβάλλουν τα ερωτήματα αυτά οι ίδιοι οι πολίτες και επομένω είναι θεμελιώδου σημασία να λάβει απαντήσεις στο Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Αλλά μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία δεν έχει γίνει δεκτή από το Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει ελπίζουμε ο διάλογος έτσι ώστε να εξευρεθεί κάποια λύση γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει χωρίς να έχει βρεθεί ε, ε, λύση σε αυτή τη δύσκολη σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπογραμμίζω στην έκθεση ότι το κυριότερο στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα. Ε, αυτός ο οποίος ε, απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει γρήγορη λύση του προβλήματός του. Ε, το 2016 έγινε αύξηση των ε, δικαστών. Έχουν βεβαίως οπωσδήποτε και τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας που είμαι βέβαιος ότι θα επιφέρουν βελτιώσεις. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε πλέον και κατευθύνες γραμμές όσον αφορά την προστασία των των καταγγελόντων. Ωστόσο υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης ε, όσον αφορά τις ε, διεργασίες ε, της δραστηριότητες των δικαστών και σε αυτές θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να είναι γνωστές οι επαφές που έχουν οι δικαστές με οποιονδήποτε. Επίσης, ο ρόλος των... Visto che questa stessa commissione ha informazioni molto marginali ε, όσον αφορά τους δικαστές εισηγητές, ε, νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη ε, διαφάνεια. Όσον αφορά δε και το ελεγκτικό συνέδριο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πλήρη πρόσβαση εις, την, εις και τις δαπάνες του δικαστηρίου. Όσον αφορά τώρα το ελεγκτικό συνέδριο, ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία και την εργασία Πρόκειται ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, ε, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά σημαντικός. Δεν έχω διαπιστώσει και δεν μπορώ επομένως να αναφερθώ σε συγκεκριμένες αδυναμίες. Απλώς θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη παρουσίαση των ετησίων εκθέσεων. Περνάω τώρα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς επίσης και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τα δύο αυτά όργανα ε, ε, έχουν πλέον προσυπογράψει συμφωνία συνεργασίας ε, για επιμερισμό των πόρων. Ζητώ όμως η χρήση των πόρων να βελτιστοποιηθεί, διότι διαπιστώνουμε ακόμα να υφίστανται επικαλύψεις όσον αφορά τα δύο αυτά όργανα που οδηγούν σε απαράδεκτη διασπάθηση χρήματος. Ε, επίσης ε, προκύπτει εδώ και το ζήτημα ε, το οποίο σχετίζεται με τις αποζημιώσεις ταξιδίου των μελών καθώς επίσης και των καταγγελόντων. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα έξοδα και οι αποζημιώσει ταξιδίου των μελών της Οικονομικής ε, ε, και Κοινωνικής ε, Επιτροπής. Εδώ θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε κάποιες μειώσεις κόστους, ίσως μέσω της χρήσης τηλεδιασκέψεων κλπ. Όσον αφορά όμως τους ε, καταγγέλλοντες, ε, ε, το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό με την Επιτροπή των Περιφερειών και ευελπιστώ ότι σύντομα θα βρεθεί λύση σε αυτήν την μακρά διαδικασία Αμφισβήτηση, ε, η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ καιρό και θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει ζητηθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών να βρεθεί λύση όσον αφορά το θέμα των καταγγελών. Τον γνωρίζω ότι τώρα υπάρχει άλλη μια υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου, ενώπιον της δικαιοσύνης δηλαδή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να λυθεί λυθεί άμεσα το ζήτημα έτσι ώστε το θέμα των καταγγελόντων να αναγνωριστεί και επομένως ε, πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μέχρι τώρα έχει υπάρξει μάλιστα και ε, ετοιμιγορία θετική. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ύπατη εκπρόσωπο για τις απαντήσεις που έδωσε στο ερευνηματολόγιο, καθώς επίσης και για το follow-up. Στην έκθεση εγώ προσπάθησα να αναδείξω ε, τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις ε, αντιπροσωπίες. Ε, έχουν υπάρξει και έχουν επιτευχθεί κάποιες πρόοδοι όσον αφορά τις κινητές μονάδες και τις μετακινήσεις. Πιστεύω πάντως ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη δυνατότητα εξοικονομήσεων κυρίως όσον αφορά ενίκεια και όσον αφορά τις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς οι διαδικασίες ε, για τις ε, συμβάσεις, τα μισθωτήρια και τα ενοικιοστάσια. Ε, θα πρέπει πάντως οπωσδήποτε να, προσπα... να γίνει προσπάθεια να μειωθεί το κόστος των των κτηρίων, ε, έστω και αν αναγνωρίζουμε ότι λόγω της ε, υψηλής παρουσίας σε πάρα πολλές χώρες ε, του εξωτερικού κάτι τέτοιο ίσως είναι δύσκολο. Βεβαίως θέλουμε να υπάρχει μια καλή εκπροσώπηση και θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων οπουδήποτε και αν δρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούν πάντως να υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την εσωτερική διαδικασία. Θα πρέπει επομένως στην Υπηρεσία Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης να βελτιωθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ε, ελέγχου, κυρίως όταν μιλάμε για μακρινές ε, χώρες. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει η μέγιστη διαφάνεια όσον αφορά την χρήση των πόρων. Τέλος, ε, ζητούμε λογικό, αποτελεσματικό και διαφανές και διαφανή προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μετακινήσεις, ακόμα και αυτές ε, ε, ε, της υπάτης εκπροσώπου. Έχουν υπάρξει πολλές πολεμικές συζητήσεις και υπάρχουν πολλές επικρίσεις όσον αφορά μετακινήσεις είτε της ιδίας υπάτης εκπροσώπου είτε άλλων μελών. Το πρόβλημα βεβαίως βγαίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Το σημαντικό είναι να υπάρξει απολογισμός και λογοδοσία όσον αφορά ε, τις δαπάνες. Ε, ολοκληρώνω ευχαριστώντας ε, την Επιτροπή μας, την Γραμματεία για την εργασία την οποία έκανε και βεβαίως περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάρκο. Θα είμαστε στους σκιώδες. Το ΕΛΚ έχει δύο σκιώδες. Η κυρία Πιτέρα, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ο κύριος Αλαφράγκα για, τους λοιπούς, ε, για τα λοιπά όργανα. Θα μας πείτε πρώτα κύριε Πτέρα εσείς για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Ναι, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Βάλη για την έκθεσή του. Την έχει δουλέψει πολύ. Έχει συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις και τα σχόλια. Θα υπογραμμίσω μόνο κάποια στοιχεία εδώ. Σημαντικά για μένα, που θα πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο συγκεκριμένα το θέμα των ανθρωπίνων πόρων, της πολιτικής για τους ανθρωπίνους πόρους και δει την ισότητα. Με συγχωρείτε για την φωνή μου, γιατί είμαι άρρωστη και την ισότητα των ευκαιριών και επίσης πληροφορίες που έχω λάβει από την ύπατη εκπρόσωπο μου δίνουν να καταλάβω ότι ανελήφθη μια σειρά δράσεων το 2016 σε επίπεδο θεσμικό αλλά και άτυπο, που στόχο έχουν να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών και έτσι να ε, εξασφαλιστεί ισότιμη ε, εκπροσώπηση των δύο φύλων και στα ηγετικά, στις ηγετικές θέσεις. Και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Επίσης ε, στις προμήθειες, στις δημόσιες αγορές χρειάζεται και εδώ μια συνεχής παρακολούθηση Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι μετά τους ελέγχους του 2016 που έδειξαν 25 περιπτώσεις όπου κάποιοι διαγωνισμοί μεγάλης, ε, μεγάλων ποσών φάνηκε να χορηγήθηκαν κατόπιν κάποιων διαδικασιών που ήγηραν ζητήματα, σαν να μην χρησιμοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες, ε, σαν να είχε υποτιμηθεί το προτινόμενο ποσό και κάποιες δράσεις θα πρέπει να αναλυφθούν, είχαμε πει τότε, για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Καλό επίσης είναι, πιστεύω, στην έκθεση. Να αναφέρουμε και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει την αποφυγή σφαλμάτων κατά την αγορά ακινήτων. Πρόκειται για μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από το 2016, αν δεν απατώμε. Και μάλιστα αυτό μετά την αμφιλεγόμενη ε, αγορά ε, ακινήτων στα Τιράνα, ακινήτου στα Τύρανα της Αλβανίας. Άρα έχουν αναλυφθεί τα σχετικά μέτρα για να αποφεύγονται τέτοιου επεισόδια στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν στοιχεία που θα χρειαστούν περαιτέρω διευκρίνηση μέσα από την έκθεση, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι δράσεις που έχουν εισαχθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας της, εξωτερικής, της υπηρεσίας της εξωτερικής δράσης. Ε, αυτά είχα να πω και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Βαλή για την πολύ καλή συνεργασία ε, για την έκθεσή του. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Sí, gracias, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Βάλε, ε, για την ε, ε, ευαισθησία που έδειξε <clears throat> έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τα σχόλιά μας στην έκθεσή του για την απαλλαγή των λοιπόν. Υπάρχει ε, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες ε, θα ήθελα να υποβάλω εν είδη και τροπολογιών. Ε, υπάρχει ένα για το οποίο δεν έχουμε νέα δυστυχώς φαίνεται ότι το Συμβούλιο για μία ακόμα χρονιά δεν θέλει, δεν δέχεται να υποβληθεί στον έλεγχο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν μας είπε κάτι σχετικό. Εάν υπάρχουν κάποιες ε, εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ε, τις παρατηρήσεις που κάνει για το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά ε, εις κάτι που με απασχολεί, ε, τα έξοδα ταξιδιού των δύο επιτροπών, Επιτροπή Περιφερειών και Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εξορθολογισμού αυτών των πολύ υψηλών από ό,τι φαίνεται δαπανών και προτείνονται κάποιες ε, γίνονται κάποιες προτάσεις για βίντεο, ας πούμε, τηλεδιασκέψεις ε, κλπ. Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε κάποιες επιπλέον ε, επεξηγήσεις σχετικά με το τόσο υψηλό ποσό των δαπανών και αν εάν μήπως μάλλον η ίδια η φύση ε, των ε, επιτροπών αυτών ε, οδηγεί σε αυτό το υψηλό ποσό ή μήπως υπάρχουν κάποιες επιπλέον προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων. Εάν εμείς γνωρίζαμε κάποια τέτοια μέτρα, ίσως θα μπορούσαμε να τα προτείνουμε θα μπορούσαμε να υποβάλουμε στα όργανα αυτά ε, τις ε, προτάσεις μας. Εάν έχετε πάντως ε, στοιχεία ε, θα μπορούσατε ίσως ε, να, μας τα, να τα υποβάλλετε ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια λογική μείωση και αποταμίευση. Γιατί κυρία, η κυρία Πιτέρα πολύ καλά εξήγησε την θέση της ομάδας μας όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εγώ νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με την πολιτική ακινήτων το πρώτο κριτήριο θα είναι η ασφάλεια. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, έχει ε, κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά συγκεκριμένες ελλείψεις και αστοχίες και είναι γεγονός ότι επί της κυρίας Μογκερίνη έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα στάνταρ και τα πρότυπα και νομίζω ότι πλέον μπορούμε και να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό ε, των ε, ε, τετραγωνικών, της επιφανίας κλπ. Αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι δυνατότητες διαχείρισης, γιατί το θέμα αυτό δεν είναι μονοσήμαντο, είναι πολύπλευρο ε, και γνωρίζουμε ότι και η Επιτροπή Εξωτερικής ε, Δράσης ε, προσπαθεί να προσαρμοστεί στις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για την εργασία του αλλά και για την ευαισθησία που έδειξε συμπεριλαμβάνοντας και τα δικά μας σχόλια στην έκθεσή του. Υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν, αλλά οπωσδήποτε ως ομάδα εμείς θα υποστηρίξουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κον. Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και να πω ότι συμφωνώ με πολλά από τα σημεία της εκθεσής του, όχι με όλα. Θα επισημάνω ένα-δύο σημεία. Περιορισμός του προσωπικού με τον κανόνα του 5% για τα όργανα. Νομίζω ότι έχει υλοποιηθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ωστόσο, έχω την επιφύλαξη ότι δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε με αυτή το καρόνα του 5% όταν μειώνεται το προσωπικό, ότι χρειάζεται και η διαδοχή, η ικανή και επαρκής διαδοχή για το μέλλον να εξασφαλιστεί. Ιδιαίτερα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης με την ενίσχυση των καθηκόντων της, και των προβλημάτων ανά τον κόσμο, θα πρέπει η δουλειά να γίνεται κατά τρόπο επαρκή, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά το υφιστάμενο προσωπικό. Για την εξωτερική υπηρεσία εξωτερική δράση είναι σημαντικό όργανο, είπαμε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις εθνικές αντιπροσωπείες γιατί στα θέματα της ε, ασφάλειας και της ενημέρωσης για την ασφάλεια πολλές φορές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της επομένω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβάλλουμε. Η ύπατη εκπρόσωπος έχει αποδείξει και επιδείξει μεγάλη διαφάνεια στην ε, λογοδοσία για τα έξοδα ταξιδιών της. Νομίζω ότι πολλοί θα μπορούσαν να τη Θετικό επίσης είναι ότι θα έχουμε στο μέλλον ε, πολύ περισσότερους μη αμοιβόμενους ασκούμενους. Επίσης ότι θα υπάρχουν προσπάθειες για βελτίωση στην πολιτική για τα κτίρια με ένα κεντρικό συντονισμό. για τον Ευρωπαίο Διαμεσολογητή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Διαφάνεια, αντιμετώπιση των προβλημάτων ή των δυσμένων συνθήκων όπως το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ε, επιθυμίες μας. Από τις 9 Νοεμβρίου υπάρχει μία πρόταση που έχει μείνει αναπάντητη του Γενικού Γραμματέα. Επομένως πρέπει να δούμε αν θα δοθεί η σχετική απαλλαγή. Η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τώρα με ό,τι επικρίσεις μπορεί να έχουμε για τα έξοδα ταξιδίων. Νομίζω ότι ορισμένα θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε ως κατηγορίες και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κύριος Αλαφράνκα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία στο παρελθόν ε, και σε θέματα ε, κοινή χρήση κτηρίων αλλά και πόρων. Η καλή συνεργασία του Κοινοβουλίου με τα δύο αυτά όργανα μπορεί να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί. γιατί έχουμε και καλή εκπροσώπηση χάρη στην Επιτροπή των Περιφερειών στις περιφέρειες, αλλά και ένα καλό εταίρο στην, ε, στο πρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Βεβαίω όλα αυτά στηρίζονται στην αμοιβαιότητα. Θα πρέπει και εμείς όταν μας ζητούν κάτι να τίνουμε ευήκον ους για το δικαστήριο. Βλέπουμε ένα σημαντικό βήμα να υλοποιείται για περισσότερη εκπροσώπηση των γυναικών. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ωστόσο. Και πάλι για το δικαστήριο για να ολοκληρώσω. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη αμοιβόμενων οσκουμένων και πάλι εδώ χρειάζεται βελτίωση. Επισημάνθη αυτό επαναλημμένος Και έχω επισημάνει και ότι το γεγονός ότι η, μια, σύντομη θητεία δικαστή μπορεί να οδηγήσει σε μια αποζημίωση, δικαίωμα σε αποζημίωση 70.000 ευρώ, μου φαίνεται υπερβολικό. Δεν μπορώ να το δεχθώ και ασφαλώς το μέλλον θα πρέπει να αποφευχθεί. Αυτά και ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από το ECR, την ALDE ή την GUE. Κύριος πράσινος. Κύριε Στάστα, είστε πάλι ο κύριο Γιάβορ. Ναι, ναι. Και θα μιλήσω αγγλικά γιατί θα διαβάσω το σημείωμα που μου έδωσε. Ο Μπένεντικτ σας ευχαριστεί για την έκθεση και θα εστιάσει σε τέσσερα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το Συμβουλίο. Γνωρίζουμε ότι έχουμε το non-paper που είχα διαπραγματευτεί εγώ για να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούν τα θεσμικά όργανα στην διαδικασία της απαλλαγής. Ορίσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής και τους ε, συντονιστές να ξεκινήσουν συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Ο Μπένεντικτ θεωρεί ότι όπως έχουν τα πράγματα αντιβαίνουν στην αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας ε, και ζητάει και από τι δύο πλευρέ ε, να προσεγγίσουν τις συνομιλίε αυτές με στόχο να επιτύχουν μια συμφωνία. Δεύτερον, ο Μπενεντίκτη θεωρεί ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο αποφασίζει για τις ευρωπαϊκές πολιτικές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο τονίζει και ο, η διαμεσολαβητής ε, στα ευρήματά της. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει να πιέζει το Κοινοβούλιο προς την πλευρά του Συμβουλίου για να σταματήσει η μυστικοπάθεια για την Επιτροπή των Περιφερειών. Μετά τις ε, δύο αποφάσεις ε, του Δικαστηρίου περί υπαλλήλων της Ένωσης ε, και τα ψήσματα του Συμβουλίου και ειδικότερα το ψήφισμα του 2015 για την απαλλαγή που καλή, καλούμε την Επιτροπή των Περιφερειών ε, να καταλήξει σε έναν δίκαιο και έντιμο συνδυασμό για τον καταγγέλλοντα. Αυτά ήταν στο προηγούμενο ψήφισμα. Βλέπουμε ότι δεν κατάφερε να λύσει την υπόθεση η Επιτροπή των Περιφερειών. Γι' αυτό οι πράσινοι θα υποβάλουν μια τροπολογία για να αναβληθεί η απαλλαγή της Επιτροπής των Περιφερειών για την έκθεση του Διαμεσολαβητή. Καλωσορίζουμε την νέα διαδικασία Fast Track για πρόσβαση στα έγγραφα των υποθέσεων. Φαίνεται ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της διαφάνειας και των εγγράφων. Υπάρχει όμως ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης από όλα τα θεσμικά όργανα. Ο Μπένεντικτ επίσης θα θέσει το πιθανό πρόβλημα των εναλλαγών αξιωμάτων και θέσεων στον διαμεσολαβητή, δηλαδή αν μετακινηθούν οι υπάλληλοι από τον διαμεσολαβητή σε μια γενική διεύθυνση η οποία είχε αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το παραθυράκι. Μετά υπάρχει το ποσοστό συμμόρφωσης με τις ε, συστάσεις που έπεσε από το 90% στο 83% και θα ζητήσει ο Μπενεντίκτ ε, από τον Διαμεσολαβητή να κάνει κάτι για να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση. Και τέλος για το δικαστήριο, ο Μπενεντίκτ θα ζητήσει μια αξιολόγηση του δικαστηρίου για τη μεγάλη εναλλαγή του προσωπικού και για το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση και οι εσωτερικέ δραστηριότητε των δικαστών. Ο Μπενεντίκτ θα ήθελε ε, τα δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να είναι δημόσια. Επίσης ε, θα ενθαρρύνει το δικαστήριο στι προσπάθειές του να μεταρρυθμίσει τους κανόνε για τη μετακίνηση του προσωπικού. Αυτά από τον Μπενεντίκτ Γιάβορο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπάρτ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει τον λόγο. Κύριε Βάλη, θα θέλατε να απαντήσετε στα σχόλια αυτά. Ναι. Ευχαριστώ, Ντέρεκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για τις ε, πολλές τους παρατηρήσεις. Χαίρομαι γιατί σε γενικές ε, γραμμές ε, επί του συνόλου των εκθέσεων έχουμε μάλλον ε, κοινή γραμμή. Θα ξεκινήσω με τη συνάδελφο Τζούλια Πιτέρα που αναφέρθηκε σε θέματα αρμοδιότητάς της για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ναι, δημόσιες, δημόσιοι διαγωνισμοί, ισότητα φύλων κτλ. Όντως αυτά πρέπει να τα δούμε και επίσης αποφυγή λαθών όσον αφορά την πολιτική ακινήτων. Πιστεύω ότι ε, τα θέματα αυτά μπορούν να μπουν ε, στην έκθεση γιατί δεν βλέπω να ε, προκαλούν προβλήματα στους άλλους σκιώδεις. Θα τα δούμε σε συνέντευξη των σκιωδών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα θέματα μπορούν να ενταχθούν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Και άλλωστε κατά αυτήν την κατεύθυνση οδηγείται και η έκθεσή μου. Όσον αφορά ε, της παρατηρήσεις του κυρίου Σαλαφράνκα για το Συμβούλιο. Απήντησε εν μέρη ο Μπάρτ γιατί ασχολείται με το θέμα αυτό. Βεβαίως, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να ανοίξει ξανά το θέμα και επομένως να το λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αναλάβει, μάλλον μας έχουν αναθέσει οι πολίτες ε, ε, αυτήν, αυτόν τον έλεγχο ε, και το Κοινοβούλιο αναθέτει τον έλεγχο στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα πρέπει να συζητήσουμε έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να ενταχθούν έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο επιτελεσματική η έκθεσή μας στο τμήμα για το Συμβούλιο. Συμφωνούμε με όσα είπατε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Όμω, Όμως όσον αφορά ε, ε, τις δαπάνες ταξιδιών ε, για την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, αυτό λέμε σχετίζεται με την φύση της δραστηριότητας των δύο επιτροπών. Όμως μιλώντας με εκπροσώπους αυτών των επιτροπών, οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν δυνατότητες εξοικονόμησης και βελτίωσης ε, με χρήση νέων τεχνολογιών ή και γιατί κάποιες ε, ε, μονοήμερες ας πούμε συνεδριάσεις ίσως θα μπορούσαν να αποφευχθούν και αντί να φέρνεις από ολόκληρη την Ευρώπη πέντε ανθρώπους ας πούμε στις Βρυξέλλες να γίνουν κάποιες τηλεδιασκέψεις ε, μας είπαν οι εκπροσώποι τους ότι είναι διατεθειμένοι να ακούσουν προτάσεις ε, και παρατηρήσεις. Και εμείς βέβαια μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτήν ε, την ευελτιστοποίηση, τον εξορθολογισμό βασιζόμενοι σε νέες τεχνολογίες και αποφεύγοντας μετακινήσεις ε, ιδιαίτερως ακριβές, δαπανηρές και όχι πάντα απαραίτητες. Όσον αφορά το συνάδελφο Κον, ε, έκανε πολύ άριθμες ε, παρατηρήσεις. Ναι, ε, βεβαίω, εάν η μείωση του 5% είναι σημαντική, πρέπει να, να υποστηριχθεί. Υπάρχουν όμως και πολλές δραστηριότητε, στις υπηρεσίες εξωτερική δράση που είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Επομένω, θα πρέπει κατά την άποψή μου να πούμε ότι ναι, είναι σημαντικό ε, να υπάρξει κάποια μείωση, ωστόσο πάντα θα πρέπει να αναλύεται σωστά η κατάσταση με τις σωστέ παραμέτρου έτσι ώστε να μην ε, ε, αποκλείσουμε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τη υπηρεσία. Επίσης όσον αφορά τις δαπάνες ταξιδίων είναι γεγονός ότι είπα ότι εκπρόσωπος είναι πολύ πιο διάφανη ε, σε, όσον αφορά ε, τις, τις ε, δαπάνες από ότι ε, άλλα θεσμικά όργανα κτλ. Αλλά ε, παρόλα αυτά βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Πρέπει να πω ότι η ύπατη εκπρόσωπος ε, ήταν εξ αρχής πάρα πολύ ανοιχτή στη συζήτηση για δαπάνες κυρίως ε, ταξιδίων αλλά υπερβολικά υψηλές. Και λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αιτιολογείται η υψηλή δαπάνη λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, επίγοντος χαρακτήρα κτλ. όταν και εφόσον υπάρχει ανάγκη ε, δεν διαφωνούμε, ωστόσο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια. Είναι γεγονό ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική έχει ε, κόστος, κοστίζει, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε το υψηλό κόστος. Όσον αφορά την ε, πολιτική ακινήτων, συμφωνούμε. Η υπηρεσία εξωτερική δράσης ε, δουλεύει, είναι παρούσα σε τρίτε χώρες, μακρινές, σε χώρες στι οποίε ενδεχομένω είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανεί, στέγη. Όμως συζητώντας και μαζί τους μου εξήγησαν ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια και εν πάση περιπτώσει οποτεδήποτε και οπουδήποτε υπάρχουν τέτοια περιθώρια ε, θα κάνουν την προσπάθεια έτσι ώστε να μειώσουν ε, το, την δαπάνη. Όσον αφορά το θέμα του Ombudsman, ε, βεβαίως θα το συζητήσουμε και με τους σκιώδεις εισηγητές γιατί κι άλλοι έκαναν, ο Μπάρτ ας πούμε, ε, τέτοιες ε, παρατηρήσεις όπως ε, αυτές τις μετακινήσεις σε άλλες θέσεις τύπου revolving doors. Σε γενικές γραμμές είναι σημαντικό να υπάρχει ισότητα ε, των φίλων όχι μονάχα στο δικαστήριο ή ε, στο ελεγκτικό συνέδριο αλλά παντού. Όσον αφορά τώρα τους ε, μαθητευόμενους, τους σταζιέρ που δεν πληρώνονται Ε, θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε αυτές οι μαθητείες, αυτές ε, οι εκπαιδεύσεις να μην κρύβουν ε, εργασία μη αμοιβόμενη. Εδώ μιλάμε για στάζ τα οποία είναι πολύ σύντομα, δεν φτάνουν ούτε στον ένα μήνα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όντως πολύ συχνά δεν υπήρχε δεν υπήρχε ε, ε, καμία αμοιβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις όντως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ε, πληρωμή τουλάχιστον αποζημίωση για τις μετακινήσεις ή για το φαγητό κλπ. Γι' αυτό λέω για να αποφύγουμε οποιαδήποτε εκμετάλλευση των νέων θα πρέπει να προβλέψουμε κάποια αποζημίωση. Έχω την εντύπωση ότι απήντησα σε όλα τα θέματα. Α, όχι, υπάρχει κάτι άλλο, ένα πολύ ευαίσθητο. Επιτροπής Περιφερειών σχετικά με τους whistleblowers, ε, τους καταγγέλλοντες. Εμείς ε, πρέπει να πω ότι ε, δώσαμε μάχη για τους πληροφοριοδότες. Εδώ έχουμε άλλωστε ετοιμιγορίες δικαστηρίων, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν έγιναν πλήρως σεβαστοί. Από όσο ξέρω πάντως, έχει ξεκινήσει και άλλη μία διαδικασία από πλευράς ε, του δικαστηρίου προς εξακρίβωση αυτής της ε, υποθέσεως. Συμφωνώ να ακολουθήσουμε σκληρή γραμμή γιατί ε, το παρελθόν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα δούμε ποια θα είναι η θέση και των άλλων, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι θα πρέπει ε, να προστατέψουμε ανθρώπους που δουλεύουν ε, στα θεσμικά όργανα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως εγώ παραμένω στην πλήρη διάθεση όλων, θα ξανασυναντηθούμε, θα ξεκαθαρίσουμε κάποια στοιχεία, ωστόσο διαπιστώ διαπιστώνω ότι γενικώ υπάρχει ε, σύγκληση απόψεων και ε, για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε συνενετική λύση, διαφορετικά λύση μέσω ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρκό. Πολλά τα θετικά σχόλια για την έκθεσή σου. Συγχαρητήρια λοιπόν. Οπότε άκουσες θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες. Η προθεσμία λοιπόν είναι 1η Μαρτίου και κλείνουμε με αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο, το υπαριθμό 60. Εγγραφή ενημέρωση για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης. ΔΕΛΤΑΠΗ μετά το 2020 ο κύριος Σάρβαμα δεν τα κατάφερε, αλλά ο κύριος, η κυρία Σμέτ συμφώνησε να τον αντικαταστήσει. ακούσουμε όμως ε, πρώτα απ' όλα το μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Γκρέκο, για το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα εγγραφό ενημέρωσης του ελεγκτικού συνεδρίου για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης η έκθεση δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και σκοπεύουμε να εκδώσουμε και άλλα τέτοια έγγραφα. Ένα για το μέλλον της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ένα για την απλοποίηση στον τομέα συνοχής και ένα για την απλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Αυτά έχουν προγραμματιστεί όλα για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και μετά αφού δημοσιευτεί και η πρόταση της Κομισιόν σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε ένα δεύτερο έγγραφο για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης και να αντιδράσουμε στην πρόταση της Κομισιόν και αργότερα στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα προετοιμάσουμε την δική μας γνωμοδότηση για την απόφαση των ιδίων πόρων που βεβαίω θα έχει σχεδιαστεί με βάση την τομιακή νομοθεσία. Συντάσσοντας αυτό το έγγραφο είχαμε μία πρόκληση το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να συμπτύξουμε 30 εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Βασιστήκαμε σε δύο γενικότερες ε, εκθέσεις του 2014. Το ένα αφορούσε την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, και το άλλο αφορούσε ακριβώς τα κενά, επικαλύψεις και προκλήσεις. Ε. Επίσης, βασιστήκαμε στις αιτήσει εκθέσεις των τελευταίων τριών ετών, 14, 15 και 16 και χρησιμοποιήσαμε και 16 ειδικέ εκθέσεις από το 2015 μέχρι 2018 και διάφορες γνωμοδοτήσεις ειδικότερα στον τομέα των ίδιων πόρων και εγκρίναμε και ένα έγγραφο ενημέρωση για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ΠΔΠ. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του περσινού ενημερωτικού εγγράφου. Βασιστήκαμε λοιπόν στον ρόλο μας στο να δίνουμε συμβουλές για το πώς δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί η διαφάνεια, η διαχείριση και η λογοδοσία από το έγγραφο της ε, Κομισιόν θα τόνιζα κάποια πράγματα. Η Κομισιόν ε, σωστά ενημερώνει τους αναγνώστες για το ότι μειώνεται από το 1,18% ο προϋπολογισμός της Ένωσης ως μέσο όρο το 93-99 σε λίγο κάτω από το 1% στις ε, τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές συμφωνούμε με τις ε, προκλήσεις ε, που αναφέρει η Κομισιόν, δηλαδή καλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες της Ένωσης ε, και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και αλληλεγγύη στην ευρωπαϊκή οικονομία και μια επιπλέον πρόκληση που αντιμετωπίζουμε από κοινού είναι το θέμα του Brexit. Και επίσης αναγνωρίζουμε ότι η προετοιμασία του επόμενου ΠΔΠ είναι κάτι το δύσκολο. Πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ υφιστάμενων πολιτικών και νέων προκλήσεων, σταθερότητας και ευελιξίας, μεταξύ των κανόνων περί δαπανών και της εστίασης στα αποτελέσματα, μεταξύ επιχορηγήσεων και άλλων μορφών χρηματοδότησης όπως η ΣΔΙΤ, και τα μεικτά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και βεβαίως ε, στην επικέντρωση σε λιγότερους τομείς. Οπότε, συμφωνούμε με τις βασικές αρχές όπως ε, τις ε, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εστιάζουμε λοιπόν σε τέσσερις από αυτές. Ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, απλοποίηση, ευελιξία και προσπαθούμε ακριβώς ε, να έχουμε αυτές τις τέσσερις αξίες σε όλα τα σημεία του κύκλου του προπολογισμού. Όταν ορίζουμε προτεραιότητες, ε, όταν εφαρμόζονται τα προγράμματα, όταν υπάρχει χρηματοδότηση και όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δικαίωση Κομισιόν προτείνει να γίνει αυτός ένας ε, βασικός στόχος του επόμενου ΠΔΠ ότι δηλαδή θα πρέπει ο κοινοτικό προπολογισμό να εστιαστεί εκεί όπου υπάρχει υψηλότερη κοινοτική προστιθέμενη αξία και αυξημένη χρήση των δημοσιονομικών μέσων και εγγυήσεων. Έχουμε παραδείγματο χάρη στα δημοσιονομικά μέσα. Κάνουμε αναφορά στην ε, έκθεσή μας 19 του 2016 όπου αναφέραμε κάποιους κινδύνους και ταυτόχρονα παραδεχτήκαμε ότι πολλοί από αυτούς τους κινδύνους ήδη έχουν αντιμετωπιστεί στην περίοδο 2014-2020. Στην πρόταση 1 βασιζόμαστε στην υφιστάμενη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την υπαρθμον 1 1-2010 και έχουμε ακριβώς την έννοια αυτή της Ευρωπαϊκής Προστομένης Αξίας που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διοργανική συμφωνίας και να ισχύει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού από τον σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή μέχρι την φάση των αποτελεσμάτων. Επίσης, συμφωνούμε με την πρόταση της ομάδας εργασίας Υψηλοπαίδου του Μάριου Μόντι για την ανάγκη να υπάρξει ακριβώς μια ανάλυση του κόστους και του ωφέλους ε, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια απλοποίηση αυτής της ετήσιας ε, έκθεσης για τα οικονομικά ωφέλη της ένταξης στην Ένωση. Στο θέμα της ευελιξίας ε, επίσης ε, συμφωνούμε με την λογική της ε, Κομισιόν ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία σε ένα σταθερό πλαίσιο. Εδώ πέρα λοιπόν βασίζουμε την πρότασή μας στο κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσης και θεωρούμε ότι τα μέσα ευελιξίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να καλύψουμε πρόβλεπτα γεγονότα και να, υπάρξει, να υπάρξουν εγγυήσεις ε, στο πλαίσιο του προπολογισμού και όχι για να αντιμετωπίσουμε τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων στα προγράμματα. Επίσης, ε, προετοιμάσουμε, κάνουμε την πρόταση να υπάρχει ένα γενικό αποθεματικό και ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο θα περιέχει κανόνες για μεταφορά κονδυλίων από τα αποθεματικά στον ετήσιο προϋπολογισμό. Μετά προτείνουμε την αναθεώρηση του ΠΔΠ και την συμπλήρωσή του με μέσο μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια τα οποία θα και την εξέλιξη διαφόρων μεταβλητών όπως την χρηματοδότηση τυχών ανοιγμάτων. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα έγγραφο το οποίο θα περιέχει ολόκληρο το συνολικό δημοσιονομικό σχέδιο το οποίο θα ενημερώνεται ετησίως με την εφαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών. Μια άλλη αρχή είναι μια προσπάθεια απλοποίησης των κανόνων με την οποία συμφωνούμε πλήρως και ήδη έχω αναφέρει τα τρία έγγραφα που θα δημοσιεύσουμε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και επίσης συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν για να απλοποιηθούν οι ήδη πόροι. Η τέταρτη πρόταση μας βασίζεται στο τρίτο κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης του 2016 και θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει η σύγκληση των προγραμματικών κύκλων για να ενισχυθεί το συνολικό τροπλαίσιο απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι είμαστε εταίροι της Κομισιόν για να αναπτυχθεί το συνολικότερο περιβάλλον απόδοσης, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με το να ευθυγραμμιστεί ο σχεδιασμός ένωσης με τους στρατηγικούς στόχους, με το να καθορίσουμε τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν, με το να μειωθούν τα προγράμματα και οι δείκτες ε, αξιολόγησης για να υπάρχουν και λιγότερες αλληλεπικαλύψεις και ένα διασφαλιστεί μια νομική βάση έτσι ώστε τα προγράμματα να έχουν μια πιο ισορροπημένη και εύκολη αναφορά για τα ζητήματα αποδοσής. Οι τελευταίες δύο προτάσεις για την λογοδοσία. Οι προτάσεις βασίζονται στην γενικότερη επισκόπηση του 2004 για τα κενά λογοδοσίας και ελέγχου θεωρούμε ότι η Κομισιόν και, από, και οι αρχές Ένωσης θα πρέπει να αναπτύξουν αρχές για την λογοδοσία και την διαφάνεια των οικονομικών της Ένωσης και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη δημοκρατική εποπτεία και γενικό κανόνα όπου αυτό επιτρέπεται από την συνθήκη θα πρέπει ε, οι φορείς να ενσωματώνονται στον κύριο προεμβολισμό της Ένωσης όπως μπορεί να γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Επίσης είδαμε τις αρχές που αναπτύξαμε το 2014 ε, υπάρχουν έξι τέτοιες υπάρχουν στο, στον πίνακα 1 μιλάμε για ξεκάθαρες ε, αρμοδιότητες, ε, δημοκρατική λογοδοσία, διαδικασίες ανάδρασης, ε, μια εντολή για ε, εξωτερικό έλεγχο και τέλος εφαρμογή των ελεγκτικών συστάσεων και παρακολούθηση των εξέλιξεων. Τελευταία πρόταση είναι να υπάρξει μια πλήρης ελεγκτική εντολή του συνεδρίου που θα και άλλους φορείς που μπορούν να εμφανιστούν όπως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και ενώ αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι αλλαγές ε, μπορεί να σημαίνουν αλλαγή της ε, συνθήκης ε, πριν γίνει αυτό εμείς καλωσορίζουμε την ευκαιρία να εκπροσωπούμαστε σε αυτούς τους φορείς, ε, στις ελεγκτικές επιτροπές. Υπάρχουν επίσης κάποια παραδείγματα ειδικών εκθέσεων όπου είχαμε δυσκολίες στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Να περάσω στην τελευταία διαφάνεια όπου βλέπετε τις προτάσεις μας που προετοιμάσαμε σε όλη την διάρκεια του προπολογισμού. Έχουμε επίσης, όπως είπα, ένα έγγραφο για τις γενικές αρχές, αλλά έχουμε και διάφορες τομεακές εκθέσεις. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για την γεωργική πολιτική έχουμε δημοσιεύσει μια σημαντική εκθέση. Για το πρασίνισμα, επίσης, μια εκθέση για τους νέους αγρότες, ε, για τους ελέγχου στην αλληλεία, ένα σημαντικό ρόλο για τους φορείς πιστοποίησης και στο θέμα της συνοχής έχουμε δημοσίευσει εκθέσεις ε, για τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό, για την ανεργία των νέων, Jaspers, ε, την διαχείριση των σειροδρομικών μεταφορών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω και μα ικανοποιούν αυτά. Πολλά από αυτά που έχουμε διζητήσει τα βλέπουμε στο κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ για το έγγραφο. Εκ μέρου του κυρίου Σαρβάμα, που είναι ο τη κυρία Σμιτ, ναι, ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ ο κύριο Σαρβάμα δεν μπορεί να είναι παρόν και με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω αναγνώσκοντα το έγγραφό του και διαβάζω στα αγγλικά. Θα ήθελα να, ευχα... να εκφράσω θερμές, θερμά συγχαρητήρια και ευγνωμοσύνη προ το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει τον θεμελιώδη του ρόλο με ένα έγγραφο ενημέρωση για τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία προτείνουν το ελεγκτικό συνέδριο για το τη προσεχή πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της επιδόσης, των επιδόσεων αλλά και τη λογοδοσία στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και όπω πολύ σωστά αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο με το έγγραφο έγγραφό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν καταστεί πιο περίπλοκα αλλά και λιγότερο συνεκτικά τα δημοσιονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ω εκ τούτου χρειάζονται εντωμεταξύ ένα νέο σύστημα δημοσιονομικό, μια νέα μεταρρύθμιση λοιπόν στον προπολογισμό η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικό και διαφανή προπολογισμό με καλύτερη στόχευση στου τομεί που εξασφαλίζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία που θα είναι πιο ευέλικτο ω προ την ε, διάθεση των πόρων εκεί όπου χρειάζονται και όταν χρειάζονται, θα είναι πιο απλό στην διαχείριση και τον έλεγχο, αλλά και πιο πρόσφορο στην λογοδοσία για τον πολίτη σε σχέση με τα ε, αποτελέσματα και τα επιτεύγματα. Πρέπει επίσης να εντοπίζονται οι ευκαιρίες για την προσθέμενη αξία από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και να αξιολογούνται οι επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών και να ε, περιορίζονται οι κίνδυνοι ή να εξασφαλίζονται εγγύησεις. Επίσης, ε, κόστος και αποτελεσματικότητα, δημοσιονομικότητα και μη της ε, συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβάλλονται μέσα από τον νέο προϋπολογισμό. Επίσης, το ελεγκτικό συνεδρίο αναφέρεται σε μια δυνατότητα για καλύτερη ανταπόκριση, μεγαλύτερη ευελιξία με ένα σύστημα αποθεμάτων το οποίο θα μπορεί να ε, καλύψει μακροπρόθεσμες δαπάνες και απρόβλεπτες εξελίξεις. Πρέπει με μεγαλύτερη έφαση να δοθεί στις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, στον Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σχεδιασμό με στρατηγικές προτεραιότητες και κύρια ε, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, περιορισμό των ε, προγραμμάτων, των δικτών και των στόχων για δαπάνες, αλλά και πιο ευθυγραμμισμένο και προσβάσιμο προϋπολογισμό όπως προτείνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Με βάση το έγγραφο, το ενημερωτικό του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά να είναι πολύ πιο διαφανή ε, με μεγαλύτερη δυνατότητα λογοδοσία να υπάρχει δυνατότητα επισκόπηση όλη τη διαδικασία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σε όργανα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού όπω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτό αυτού όπω Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει παρησία και λογική και αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα να τα λάβει υπόψη κατά την κατάρτιση των προτάσεων για το Πουδουπού. Το ελεγκτικό συνέδριο υπογραμμίζει πολύ σημαντικά στοιχεία και σημεία και δίνει τα κλειδιά της επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σωστά επισημαίνεται η ανάγκη για τον προγραμματισμό των δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο προσεκτικό με την δυνατότητα για διαχείριση, παρακολούθηση, ε, αξιολόγηση με πιο αποτελεσματικό, απλό και διαφανή τρόπο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών. Τονίζουμε λοιπόν τη σημασία αυτή τη έκθεση και των προτάσεών τη και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι περιλάβει προσοχή προτάσει για το Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κυρία Κλαπαϊό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ καλά προετοιμασμένη ενημέρωση. Συμφωνώ απολύτως ε, με τις πολύ καλές προτάσεις σας, ε, τις οποίες ε, συμμερίζομαι. Θα ήθελα μόνο να υποβάλω κάποια ερωτήματα, ίσως πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να τα αναφέρουμε. Στο Reflection Paper αναφέρεται ότι ε, στο νέο πολιτές ε, ε, πρόγραμμα θα πρέπει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να αποτελέσει κύριο κριτήριο και ότι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν καλύτερα, καλύτερες επενδύσεις. Αυτό θα βεβαίως σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερο κλίμα. <laughs> Α, να τα λέω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, έλεγα ότι ε, υπάρχουν ε, άμεσες και έμεσες ε, αιτίε για τις οποίες μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και δεν εξαρτώνται όλες από τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα, ίσως δυσεπίλη το άλλο να θα συζητήσουμε μαζί, πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς με μία μόνο φράση την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία σε έναν πολίτη. Γιατί νομίζω ότι ε, ε, εάν η εξήγηση και ο ορισμός είναι απλή, τότε είναι, θα είναι πολύ θετικό όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους μελλοντικούς παίχτες ε, της ευρωπαϊκής ε, χρηματοδότησης. Επίσης γίνεται λόγο σε με περαιτέρω χρήση των δημοσιονομικών ε, εργαλείων αλλά εδώ τα διλήμματα είναι διπλά. Πρώτον, από την άποψη των δημοσίων οντοτήτων, όπως ας πούμε δήμοι, κοινότητες κλπ, που δεν ελκύονται ιδιαίτερως από τα χρηματοδοτικά, χρηματοπιστωτικά εργαλεία ε, και ε, επίσης ε, εκεί παίζει και διαφορετικά η επεξήγηση που δίνει κανείς στις κρατικές επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις. Το δεύτερο δίλημα αφορά τα δάνεια, grants. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιος κατά την άποψή σας είναι ο ρόλος των χρηματοδοτικών εγγυήσεων και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρετε ότι η αρχή της επικουρικότητας και της απλούστευσης δεν είναι είναι πάντα ε, ε, παρόν, παρούσες ε, ταυτοχρόνως, δεν πάνε χέρι με χέρι στις δημόσιες προμήθειας. Υπάρχουν 28 επιμέρους ειδικέ ρυθμίσεις για την ε, υλοποίηση του ιδίου ε, νομοθετήματος. Ποια είναι η άποψή σας ε, από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου, από πλευράς του ελέγχου. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η απλούστευση. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα απλουστευμένο περιβάλλον και αν ναι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θέλω να σας δώσω το λόγο κύριε Γκρέγορ και μετά να ακούσουμε την Επιτροπή. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ευμενή σχόλια, για το ενημερωτικό υπόμνημα και τις ε, σχετικές ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στις τρεις αυτές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Προσταμενή Αξία. Πιστεύω ότι ο ορισμός που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση για το 2011 είναι αρκετά απλός και προ... την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία από την παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με αυτό το οποίο θα είχαν επιτύχει τα κράτη-μέλη ε, παρεμβαίνοντας ε, μόνα τους. Βεβαίω αυτό είναι πολύ πιο απλό από ό,τι θα μπορούσε κανείς να περιγράψει. Είχαμε το 2017 ένα σχεδιασμό μιας ε, ομάδας εργασίας, ομάδας ποιότητας που θεσπίστηκε προκειμένου να αξιολογήσει και να περιγράψει τη δική μας θέση, τις δικές μας θέσεις για την προσθεμένη αξία. Είναι στη δουλειά ήδη και πολύ ευχαριστώ να συμπεριλάβουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις σχέσεις, στις ιδέες μας. Αλλά βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την ε, πολιτική έως το 2020. Θα περιλάβουμε λοιπόν θέματα προσθέμενης αξίες για το δημοσιονομικό μέσο. Καταγράφω τις προτάσεις, αναφέρομαι σε μια ειδική έκθεση 2016 που ονομάζεται ειδική έκθεση για τα χρυσά ταμεία όπως την έχουν πει Εκεί έχουμε προσπαθήσει να επισημάνουμε κάποιους κινδύνους από την αξιοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων που ιδίως αφορά ε, χρηματοοικονομικά μέσα στη διάθεση των κρατών μελών. Και γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με το αν πρόκειται για, ευρωπαϊκό, για εθνικό επίπεδο ή κεντρικό επίπεδο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λοιπά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως ε, καλούμε τον καθαρά να δείξει την απαραίτητη σύνεση, φρόνηση κατά την ε, διατύπωση των προτάσεων. Επίσης πιστεύω ότι είναι καλό να επικεντρωνόμαστε στις δημόσιες δαπάνες όταν κάνουμε αυτή την για, την, ε, για τον εξοραϊσμό των δαπανών. Είναι εύκολες οι ε, επικρίσεις αυτές από τα κράτη-μέλη, αλλά εγώ θα επιμείνω στις δικές μου και προσωπικές θέσεις τι ήταν αυτό που χαρακτήρισε το φαινόμενο αυτό, πώς προκύπτει. Μπορεί και το ελεκτικό συνέδριο να έχει κάποιο ρόλο, γιατί μπορεί κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις μας στο παρελθόν να οδήγησαν τα κράτη-μέλη σε διαμόρφωση συστημάτων πιο περίπλοκων, λιγότερο διαφανών. Ευπρόσδεκτες πάντως οι προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση των κανόνων. Με ένα εγχειρίδιο οδηγό για του διάφορους τομείς. Δημόσιες προμήθειες. Θα ήταν επαναστατικό αυτό βέβαια. αλλά καθώ τα συστήματα διαχείρισης των δημοσιονομικών και των ελέγχων βεβαίων των, των, των δαπανών παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε αυτή την πορεία, αυτή την εξέλιξη για τις δημόσιες προμήθειες. Και πρέπει να δεχθούμε κάποιε συνέπειε για τις ε, εθνικές ένωμες τάξεις. Βεβαίως, μπορεί να απλουστευθεί ιδιαίτερα η δουλειά των ε, δικαιούχων, των αλλά από την άλλη δεν θα τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Ή ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διτηρούν τον έλεγχο αυτών των δαπανών. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. να διατηρουν τον ελεγχο Πρέζα, Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, πω ότι μπορώ να συμφωνήσω με το έγγραφο της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, καθότι διαπιστώνεται υψηλός βαθμός ε, σύγκλησης με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο Reflection Paper για το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται εστίαση στην ευρωπαϊκή και νέα προστιθέμενη αξία, στην ε, αντιδραστικότητα, στην ε, ε, θέση αρμοδιοτήτων σε, συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένα πεδία, θέμα το οποίο σημειώθηκε επανειλημμένα. Και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει λοιπόν σύγκληση απόψεων όσον αφορά κοινού στόχου Εντάχει θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα τα οποία έδειξε ο κύριος Γκρέγκορ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο ε, είναι η αδελφή, ας πούμε, ή ο αντικατοπτρισμός της επικουρικότητας. και θα πρέπει να χρηματοδοτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η παρούσα μέτρηση δεν είναι τόσο άμεση ε, όσο φαίνεται να αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο. Και βεβαίως ε, δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε, μετρά, οτιδήποτε είναι μετρήσιμο πρέπει να μετρηθεί, αλλά οτιδήποτε είναι σημαντικό προσμετράται. Πάντως ε, πρέπει να εστιάσουμε ε, στο να δείξουμε την πραγματική θέμενη αξία και να ε, επιμείνουμε ε, στα επιτεύγματα αλλά και σε άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι τόσο μετρήσιμα. Ας πούμε, το, ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων μπορεί να μην είναι απόλυτα μετρήσιμος αλλά οπωσδήποτε δίνει θετικές θεωρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ευελιξία, η Κομισιόν μπορεί να συμφωνήσει με τις κεντρικές προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι προτάσεις για το επόμενο ε, πι δελτα πι ε, μπορεί να είναι πολύ σωστές. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να δοθούν ε, στα εργαλεία έτσι ώστε να επιτρέψουν πιο ευέλικτη χρήση των κονδυλίων εντός των κεφαλαίων αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο επόμενο ΠΔΠ. Η Κομισιόν ε, δεν, ε, δεν κάνει αξιολογήσεις βάσει των net balances ε, τόσο εύκολα. Δεν συμφωνεί απολύτως με μια τέτοια αντιμετώπιση. Πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν υπολογισμοί βεβαίως και θα πρέπει να γίνουν και οι, οι διάφορες εξισώσεις. Ε, ε, εμείς και για το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουμε ευρύτερη ε, προσέγγιση σε μια προσπάθεια να συνυπολογίσουμε και τα στοιχεία τα οποία εκφεύγουν του απλού λογιστικού, της απλής λογιστικής θεώρησης. Επίσης, όπως και πρόσφατα για την ενδιάμεση επισκόπηση, ε, έτσι και τώρα ε, για τον και για τον αναθεωρημένο ε, δημοσιονομικό εργαλείο, ε, Βεβαίω ε, συζητιέται το θέμα και στι ε, συζητήσει. Υπάρχει άρθρο του άρθρου 146, βάσει του οποίου η ε, Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία σειρά καλά πιστοποιημένων ε, ε, προτάσεων και αιτιολογήσεων των κινήσεων της ε, έτσι ώστε να μπορούν να δικαιολογηθούν και οι δαπάνες πληρωμών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω ότι επί της ουσίας ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχει μεγάλο βαθμό σύγκληση. Όσον αφορά την απλούστευση πιστεύω ότι ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια απλούστευσης ε, με τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και υπάρχει επίσης και μεγαλύτερη ευελιξία. Οπωσδήποτε η πρόταση του ελεκτικού συνεδρίου για μείωση του αριθμού ε, των ε, προγραμμάτων είναι μια ε, πρόταση την οποία θα, η οποία θα ληφθεί υπόψη και θα γίνει μια προσπάθεια υλοποίησής της. Όσον αφορά την λογοδοσία, η Κομισιόν φρονεί πως η λογοδοσία παρέχεται ε, μέσα από όλο το σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού ε, και μέσω των ε, δημοσιονομικών εργαλείων όσον αφορά μάλλον τα εργαλεία δημοσιονομικά τα οποία είναι εξωτερικά της Κομισιόν, υπάρχει και σε αυτά αντίστοιχος έλεγχος. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Ζαμπάγεβα σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δημοσιονομικά εργαλεία, αν χρησιμοποιούνται μόνο, είναι καλά, κατάλληλα μόνο ε, για τον ιδιωτικό τομέα ή και για το δημόσιο. Ε, οι εγγύησει προϋπολογισμού και τα δημοσιονομικά εργαλεία έχουν έννοια ε, για, πρόγραμμα, για προγράμματα από τα οποία ευελπιστούμε, προσδοκούμε ε, μελλοντικές ε, ε, ροές ανταπόδοσης. Όταν έχουμε προγράμματα όπως ας πούμε είναι προγράμματα στέγασης που θα πληρωθούν ας πούμε από το εισόδημα μέσω φόρων ή μέσω άλλου δημοσίου εισοδήματος, ναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ας πούμε για να ε, χρηματοδοτηθεί να χρηματοδοτηθούν ε, προγράμματα συνεργασίας ιδιωτικού δημόσιου τομέα ε, έτσι ώστε να μειωθεί το επίπεδο κινδύνου, να αυξηθεί η ελκυστικότητα και έτσι ώστε να προσελκυθούν φορείς οι οποίοι δεν θα προσελκύονται διαφορετικά. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη μόχλευση των χρημάτων ε, που λαμβάνονται από τον φορολογούμενο και εν τέλει μπορούν να βελτιώσουν την τελική αξία του χρηματοδοτούμενου αντικειμένου. Τέλος, όσον αφορά την λογοδοσία η οποία ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σημειώνω ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ε, λάβει χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Επομένως, ε, θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες μεταξύ δικαστηρίου και άλλων ε, οργανισμών. ούτε ή άλλως οι υποχρεώσεις ε, καταγράφονται ε, ρητά ε, στους κανονισμούς και επομένως δυσκολευόμαστε να δούμε πώς μπορούν να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις. Τέλος, γενικά για το briefing paper, βεβαίως πρόκειται ε, για ε, ένα πολύ ε, πολύτιμο επιπλέον στοιχείο, τροφή για σκέψη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, διαβάζοντάς το βεβαίως, κάπου τα έχουμε ξαναδεί αυτά και το ερώτημα είναι πώς θα τα εφαρμόσουμε και δεν είμαι σίγουρος αν τα έχω αντιληφθεί όλα σωστά. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση. Το θέμα δηλαδή της προσαρμογής των κύκλων είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Το θέμα της λογοδοσίας, το να καλύψουμε τα διάφορα κενά. Θέλει η συγγήτρια πάλι τον λόγο, η κυρία Σμιτ. Όχι. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εντυπωσιακή δουλειά και αναμένουμε και τις υπόλοιπες ε, συνεισφορές. Ε, εγώ αναμένω δε το μέλλον της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε περνάμε τώρα στο σημείο 61 της ημερήσιας διάταξης η ειδική έκθεση για το πρασίνισμα. του ελεκτικού συνεδρίου είχαμε ήδη μία σύντομη παρουσίαση και συμφωνήσαμε να γίνει μία πλήρης παρουσίαση της έκθεσης. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας πείτε τα όσα δεν ξέρουμε. Η συγητής είναι ο συνέλφος Τεχόφσκι ε, Νομίζω και οι σκιώδεις συγητές είναι εδώ. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τα ευρήματα της έκθεσης για το πρασίνισμα που είναι ένα πιο περίπλοκο σύστημα στήριξης του εισοδήματος. Ε, πρασίνισμα ξεκίνησε ως ένας τύπο, νέος τύπος άμεσων πληρωμών προς τους αγρότες το 2013 για να ανταμυφθούν οι αγρότες για τα δημόσια αγαθά που παρέχουν και να ενισχυθεί έτσι η περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση της ΚΑΠ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει 12 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος στο πρασίνισμα, δηλαδή 30% όλων των άμεσων πληρωμών της ε, γεωργικής πολιτικής και 8% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι αγρότες λαμβάνουν, έλαβαν τις πρώτες ε, τέτοιες πληρωμές ε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 για αιτήματα που υπέβαλαν το 2015. Τα βασικά λοιπόν ευρήματα του ελέγχου είναι ότι όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή το πρασίνισμα θα έχει μικρή επίδραση στην ε, κλιματική απόδοση της ΚΑΠ καθώς οι απαιτήσει δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες και λόγω των πολλών εξαιρέσεων πολλοί αγρότες, γύρω στο 65% αυτών μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση χωρίς να έχουν κάποιες ιδιαίτερες υποχρεώσεις. Οπότε έχουμε πολύ περιορισμένες άλλαγες ε, γύρω στο, 50, στο 5% της ευρωπαϊκής καλλιεργήσιμης γης. Να αναφερθώ τώρα στο νούμερο το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 73% των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων έχουν τουλάχιστον μία υποχρέωση πρασινίσματος. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως ακόμα και εάν ε, υπάρχει υποχρέωση για ένα εκτάριο από τα 100 εκτάρια ενός αγροκτήματος, η Κομισιόν μετράει και τα 100 εκτάρια. Ακόμα και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην πρακτική που ακολουθούσε ο αγρότης, γιατί ακολουθούσε κάποια παρόμοια πρακτική από πριν. Οπότε αυτό δεν θα αλλάξει ακόμα και αν καλύπτουν 3, 5 ή και μεγαλύτερο ποσοστό της 100 της καλλιεργήσιμης γης. Οπότε θεωρούμε ότι ο δείκτης αυτός ε, έχει περιορισμένη χρήση για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα του πρασινίσματος. Βρήκαμε ότι η Κομισιόν δεν έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους ή δεν έχει καθορίσει το τι θα πρέπει να πετύχει το πρασίνισμα για το περιβάλλον και το κλίμα και δεν δικαιολογείται από το περιβαλλοντικό περιεχόμενο της πληρωμής. Ε, κατά κανόνα οι πληρωμές είναι γύρω στα 80 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ η Κομισιόν υπολογίζει πως το μέσο κόστος ε, δεν θα υπερεύαινε τα 30 ευρώ. Η μελέτη λοιπόν του Κοινού Κέντρου Έρευνας δείχνει πως ε, έχουμε διαφορετικό αντίκτυπο, δηλαδή λιγότερο από 10 ευρώ για τους περισσότερους αγρότες, ενώ πάνω από 100 ευρώ για ένα 2 των αγροτών. Οι περιορισμοί στον σχεδιασμό μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ε, πρακτικών αυτών. Η φορά δεν ε, μπορεί να ε, έχει τα ίδια αποτελέσματα με την αλλαγή των καλλιεργειών και Βεβαίω το ότι κυρίως εστιαζόμαστε σε περιοχές ε, οικολογικής ε, εστίασης σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη επίδραση στην βιοπικιλότητα. Το πρασίνισμα έχει προσθέσει σημαντική πολυπλοκότητα στην ΚΑΠ που δεν δικαιολογείται από τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει. Η πολυπλοκότητα αυτή προκύπτει από τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ πρασινίσματος και άλλων περιβαλλοντικών μέσων της ΚΑΠ, μεταξύ των οποίων οι ορθές ε, περιβαλλοντικές ε, συνθήκες και τα κράτη-μέλη δεν εκτιμούν την πολυπλοκότητα αυτή καθώς αφορά ειδικά τον ορισμό περιοχών οικολογικής εστίασης για να μεγιστοποιηθεί ακριβώς ε, το όφελος. Ε, αντιθέτως προσπαθούν να εφαρμόσουν το πρασίνισμα με έναν τρόπο που θα επιβαρύνει λιγότερο τα ίδια και τους αγρότες. Με βάση αυτά τα ευρήματα κάνουμε τις εξής συστάσεις για την επόμενη μεταρρυθμίση της ΚΑΠ. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναπτύξει μια πλήρη λογική παρέμβαση ε, για την συνεισφορά της ΚΑΠ στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθήσει τις αρχές ότι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση στις πληρωμές της ΚΑΠ μόνο εάν ανταποκρίνονται σε κάποιες βασικές περιβαλλοντικές διατάξεις που καλύπτονται από τις τωρινές διατάξεις και το, πρασίνισμα, ότι ειδικέ και τοπικές ε, και κλιματικές ανάγκες ε, θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ισχυρότερων προγραμματισμένων δράσεων, να ανταμείβουν τους αγρότες για τις υπηρεσίε τους που υπερβαίνουν τις βασικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και πω τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποδεικνύουν πως έχουν επιλέξει επιλογέ, οι οποίε είναι αποτελεσματικέ σε σχέση με την επίτευξη των στόχων. Σα ευχαριστώ. Πολύ σημαντική ειδική έκθεση, θα πρέπει να την ξαναδούμε βεβαίω ε, και παραμένουν τα ερωτηματικά μα. Σε σχέση με τι σχετικά περίφραστε επικρίσει με πόρνα το κύριο Τσεχόφσκι είναι ο εισηγητή και θα του δώσω το λόγο αμέσω. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βέβαια δεν τηρούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα όπως το είχαμε προβλέψει, αλλά έχω μάθει να προσαρμόζομαι. Ελπίζω να μην ε, έχασα τίποτα σημαντικό την ώρα που απουσίαζα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη σημαντική έκθεση και νομίζω ότι μας δείχνει ακριβώς το λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ, γιατί κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας πολιτικός, πολύ σημαντικός πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής και μας δείχνει τη σημασία της κοινή γεωργικής πολιτικής που ταυτόχρονα όμως απαιτεί και μια διεξοδική α, μεταμόρφωση, μεταρρύθμιση. Έχουμε το πρασίνισμα κατά σημαντικό ποσοστό 8%. Βέβαια βλέπουμε με, με ανησυχία τις ε, διαπιστώσεις τις σχετικές για το κομμάτι αυτό γιατί βλέπουμε ότι δεν προχωρεί όπως θα έπρεπε στα αποτελέσματα που είχαμε αρχικά επιδιώξει. Οι αρχικές προσδοκίες σε σχέση με το πρασένισμα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό κανονικές συνθήκες ε, υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν σαν στόχο την ε, μείωση των ε, συνεπειών στην κλιματική αλλαγή από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εδώ όμως αυτό δεν εξασφαλίζεται και πρέπει να γίνει εκβάθρων μεταρρύθμιση του προγράμματος, αλλιώ να μπει ένα τέρμα. Είναι με περισσότερο από ό,τι χρειάζεται το πρασίνισμα και πιστεύω ότι η λογική του εργαλείου αυτού δεν υπηρετείται επαρκώς. Πιστεύω ότι είναι πολύ περίπλοκο το μέσον δεν έχει αρκετή διαφάνεια, εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους και δι καταχρήσεις και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του ελεγκτικού συνεδρίου είναι εκτεθειμένο σε πολλές ε, παραβιάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της ε, καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής αλλά με πιο αποτελεσματικά μέσα. Αυτό προσπαθώ να πω εγώ στην έκθεσή μου. Το πρασίνισμα πρέπει να εξεταστεί μέσα στις μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, βεβαίως θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει για το αν είναι σκόπιμο να ε, μειώσει ενδεχομένως ε, την υποστήριξη της ενισχύσης που προσφέρονται για το greening, για το πρασίνισμα ή αν θα πρέπει να αξιοποιηθούν διαφορετικά μέσα που ενδεχομένως να υπηρετούν καλύτερα το στόχο της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντενμπαχ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ θερμά και εγώ το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και τον κύριο Τόμας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και το βλέπουμε γιατί την ξανασυζητούμε. Είμαστε σε μια ε, επικαιρότητα καυτή. Πρέπει να συζητήσουμε και την κοινή γεωργική πολιτική. Βεβαίω έρχεται με μια κάποια καθυστέρηση δυστυχώ στην όλη αυτή διαδικασία η έκθεση, γιατί θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν προτιμότερο να είχαμε νωρίτερα κάποιες ιδέες και προτάσεις για μια αλλαγή νοοτροπίας και σχεδιασμού. Ε, ανέφερε ήδη ο κύριος Τσεχόφσκι τα σημαντικά από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει για την κοινή γεωρική πολιτική φιλόδοξα σχέδια. Ε, παραδείγματι για το greening του πρασίνισμα, την οικολογική προσέγγιση. Είχε κάνει προσδιορισμό των στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ωστόσο να δώσει μια συγκεκριμένη εστίαση σε αυτούς τους στόχους. Το επικρίνει άλλωστε και το ελεκτικό συνεδρίο. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι έχουν ε, τα ουσιώδη αυτά μέσα για την υλοποίηση του ε, στόχου αυτού υπονομευθεί, υποβαθμιστεί, καθώς εισάγονται από τα κράτη-μέλη κάποια συστατικά στο σύστημα, τα οποία παρεμβαίνουν σε πολύ έντονο βαθμό. Και ενώ θα έπρεπε να υπηρετείται η περιβαλλοντική πολιτική, το μέσον αυτό μετατρέπεται σε ένα ε, μέσον ενίσχυσης του εισοδήματος των γεωργών. Στο πεδίο αυτό λοιπόν και χωρίς να θέλω να αφαιρέσω ούτε δεκάρα από κάποιον γεωργό Ευρωπαίο, ε, πρέπει να δούμε εάν τηρείται ο στόχος, εάν υπηρετείται όπως τον έχουμε προβλέψει και αντίστοιχα για το μέλλον πρέπει να δώσουμε σαφείς ορισμούς του στόχου αυτού πιστεύω. Αυτό ήταν και η λογική της ε, τοποθέτησης σήμερα της παρέμβασης όπως υπόθηκε. Αυτό που θα ήθελα να αποφύγουμε ωστόσο θα ήταν ε, από τη συζήτηση να προκύψει το συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόμαστε την οικολογική προσέγγιση, του πρασίνισμα και έτσι κάνουμε και τη σχετική οικονομία σε πόρους. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ανάγκη για οικολογική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε ακόμη και πάντα πράσινη γεωργία, αλλά με συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένα καθήκοντα και ταυτόχρονα για τα κράτη-μέλη, τα οποία βεβαίως αναλογώς και της γεωγραφικής ε, θέσεως ή των προκλήσεων που μπορούν να αντιμετωπίζουν και είναι διαφορετικές πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το καθένα από αυτά, χρειάζονται μια διαφορετική, μια ευελιξία σημαντική. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει αυτή η ευελιξία να επιτρέπει να ε, καταλήγουν σε διαφορετικές ε, λύσεις που, παραμένουν αδιαφανείς, δηλαδή να υψώνονται τείχη αδιαφάνειας, γιατί δεν είναι πολλές φορές δυνατόν από αυτά που βλέπουμε μέσα από ένα ευρύ φάσμα που ναι εντάξει πρέπει να υπάρχει η ευελιξία, αλλά από το ευρύ αυτό φάσμα μέσων που έχουν του τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να προκύψει αυθαιρεσία ή αδιαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ και τη Γεωργική Επιτροπή για την έκθεση αυτή, συζητείτε εγκαίρως και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να συμβάλλουν οι συνάδελφοι της, Επιτροπή της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό, είναι πλέον αρμόδιοι για το πρασίρισμα, το οποίο όμως πρέπει να υπηρετεί τους στόχους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνεται. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιλαμπάιουα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να συμφωνήσω ότι τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και του ε, εισηγητού είναι ότι το, το πρασίνισμα δεν θα δώσει τελική λύση για το κλίμα. Ίσως και σε σχέση και με αυτά που είπε η Σάρφος Καρίν προηγουμένως νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Ε, εγώ έχω δύο ερωτήματα, ε, μία στο, για την Κομισιόν, μία για το ε, ε, ε, Ελληνικό συνέδριο, σημείο 28 της έκθεσης, αναφέρει σε περίπτωση διαφοροποίησης των, των καλλιεργειών, τότε θα πρέπει να εισαχθεί το πρασίνημα χωρίς καμία αλλαγή στις καλλιεργητικές συνήθειες. Αυτό γιατί έχουν ήδη καλυφθεί οι στόχοι του πρασινίσματος την προηγούμενη χρονιά, είτε γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα πράγματα. Οι νέοι γεωργοί οι οποίοι θίγονται ε, από, τις, από τους νέους ε, ε, κανόνες είναι 1% και όσον αφορά το, την οικολογική εστίαση το ποσοστό ανεβαίνει περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη χρηματοδότηση της Κομισιόν και ποιες είναι οι προσδοκίες Κομισιόν ε, οι προσδοκίες σας, προσδοκίες αντικτύπου όταν καθορίζεται το πρασίνισμα, αναφέρομαι σε σύνολο καλλιεργημένης γης. Και ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, που ε, θα μπορούσε να θεωρηθεί από το ελεγκτικό συνέδριο ως σημαντικός ή και επιτυχής. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν άκουσα την παρουσίαση Πάντως το ζήτημα του προσυνείσματος ε, είναι ότι οργανώθηκε με τρόπο που άφησε άφωνους ε, περίπου τους ανθρώπους. Το θέμα ε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε αυτό στη χώρα μου ήταν απίστευτος και το γεγονός ότι μειώνονται και τα χρήματα που δίνονται στη γεωργία δεν βελτιώνει την ε, ε, κατάσταση. Όσο πιο ψηλές ιστορικές, ε, ιστορικά επιδοτήσεις έχει πάρει κανείς, τότε και το πρασίνισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος από βασικές πληρωμές παίρνει 40 ένα εκτάριο θα έχει 20 για το πρασίνισμα. Ε, και ε, σε βασικές ε, πληρωμές μπορεί να φτάσουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο γειτονικές καλλιεργημένες περιφέρειες και δύο γειτονικούς γεωργούς. Ε, αυτό είναι αστείο. Ο τρόπος δηλαδή που έχει οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα είναι αστείο. Ε, είναι κρίμα βέβαια γιατί υπήρχε μεγάλο δυναμικό και αυτά που θέλαμε, η βιωσιμότητα που θέλαμε να επιτύχουμε ε, με το πρασίνισμα, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεν, ε, ε δεν γιατί δεν επιτέχανεται ε, πολέμηση πολιτικής της ε, κλιματικής αλλαγής αν δώσει σε ένα γεωργό 500 ευρώ και σε το διπλανό γεωργό 20. Ευχαριστώ. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, θέση βέβαια. Από τη Γενική Διεύθυνση για τα Γεωργικά Θέματα έχουμε την υποστήριξη κύριε Πάσκου Προ του γεωργού, Θα μας απαντήσετε, δεν γίνεται κάθε χρόνο να δίνουμε 5 δις ευρώ χωρίς αποτελέσματα χωρί Γιατί αυτό μας λέει η ειδική έκθεση. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι όπως έχει τώρα η κοινή γεωργική πολιτική. Η Επιτροπή τι προτείνει. Ή μας λέτε να κανουμε ετσι οπως εχει τωρα η κοινη πολιτικη η επιτροπη τι προτεινει η μα λετε να προχωράει το σύστημα, να τρέχει μέχρι ότου γίνει μεταρρύθμιση. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό συμβει αυτο βεβαίω. Άρα, τι προτείνει η Επιτροπή τώρα. Δεύτερο και ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο. Έχουμε στον πίνακα τρία, μείωση του επιδιωκόμενου επίπεδου πρασινίσματος κατά την νομοθετική διαδικασία. Ενδιαφέρον. Στο τρίτο, στην τρίτη εικόνα. Η επικόνηση. Γιατί δείχνει και τους κινδύνους από την δημοκρατία. Ο δρόμο προς την κόλαση είναι στρωμένο με καλές προθέσεις. Τι θα πούμε λοιπόν όταν έρθει η ώρα να εξηγήσουμε ότι κάποιοι υποφελήθησαν, ε, αποκόμισαν ίδιον όφελος από όλη αυτή την ιστορία. Ή έχουν, εν πάση περιπτώσει, μόνοι τους ε, ε να αποφασίζουν. Έχουν και το πεπόνι και το καρπούζι τους και το μαχαίρι του επίν. Επομένως λοιπόν πώς θα αποφύγουμε τα προβλήματα στο μέλλον, προβλήματα που τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Και ε, ευχαριστώ ε, με την επιτάσσεως στο ελεγκτικό συνέδριο, γιατί ε, βεβαίως και εμείς τα είχαμε το πίστηφλοι, δεν είμαστε. Αλλά είχαμε δει και μας επιδεικνύει, μας αποδεικνύει το ηλεκτρικό συνέδριο ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα μπροστά μας. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Το να μην κάνουμε τίποτα αποκλείεται. Για να δούμε όμως ο κύριος Στάστη έχει να πει συνάδελφος Στάς. Ναι, δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά ακούγοντας όλους τους ε, συναδέλφους ε, θυμάμαι όταν είχαμε κάνει τη μεταρρύθμιση της γεωργικης πολιτικης πολιτικής 2012-2013 και έχω την εντύπωση ότι η αρχική πρόταση του Επιτρόπου Τσιόλος ε, τότε προέκυψε από την συζήτηση και πρέπει νομίζω να κοιτάξουμε στον καθρέφτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας ε, συνεισέφεραν στο εξασθένισμα της ε, πρότασης της Κομισιόν και τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα του ελεγκτικού συνεδρίου ότι τα μέτρα πρασινίσματος όπως τα περιγράφει η νομοθεσία δεν ε, λειτουργούν. Βεβαίω ήταν πολύ καλύτερες οι αρχικές προτάσεις ε, του Επιτρόπου Τσιόλος από αυτό στο οποίο καταλήξαμε και το ερώτημα προς την Κομισιόν είναι όταν θα φέρει τις νέες ε, προτάσεις για τη μεταρρύθμιση, πότε θα είναι Μάιο, Ιούνιο, αν θα έχουν κάποια ουσία πρασινίσματος και αν θα βασίζονται στις αρχικές προτάσεις του Επιτρόπου ε, Τσιόλος. Αυτά έτσι στο περιθώριο της συζήτησης. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχει κάποιος ε, χρόνο να πάει στην ε, Επιτροπή Γεωργίας. Ναι, η κυρία Κάνιμπαχ. Ε, πρέπει να το παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι. Ναι, ο εισηγητής εδώ πέρα της απαλλαγής ε, μας κοιτάει. Ναι, θα πρέπει νομίζω να το δούμε κάπως πιο σοβαρά. Ίσως θα μπορούσε να στείλει κάποιον η γραμματεία, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, κύριε Πάσκο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής. Να σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές δηλώσεις για την άποψή μας όσον αφορά την έκθεση και μετά θα επανέλθω σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα τα οποία ετέθησαν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως ε, η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την ειδική έκθεση. Νομίζω ότι το πρασίνισμα ήταν η βασική καινοτομία της προηγούμενης μεταρρυθμίσης και είναι σημαντική, αν και είναι δύσκολο όταν μιλάμε για περιβαλλοντική πολιτική, να αξιολογήσουμε ήδη την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής. Αλλά θα ήθελα να πω πως η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την έκθεση η ουσία όλων των συστάσεων είναι αποδεκτή από την Κομισιόν και βεβαίως ε, όταν θα έχουμε μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική για την περίοδο μετά το 2020 το ελεγκτικό συνείδριο τόνισε κάποιες αδυναμίες ε, και Βεβαίω συμφωνούμε με αρκετές από αυτές αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάποια ερωτήματα, ευρήματα μας συγχωρείτε, του ενεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική απόδοση της πολιτικής. Πρώτα απ' όλα, το ενεκτικό συνέδριο υπενθυμίζει την άποψη της Κομισιόν ότι το πρασίνισμα έχει την δυνατότητα, δυνατότητα υπενθυμίζω, να συνεισφέρει πριν από την εισαγωγή του το 2015 και ότι το 5% της ευρωπαϊκής καλλιεργήσιμης γης ε, υφίσταται και καλύπτεται από κάποια σχετική υποχρέωση και αρχικά βέβαια αυτό το ποσοστό θα ήταν ακόμα υψηλότερο αλλά βέβαια ε, εισήχθησαν πολλές ε, εξαιρέσεις και η πλειοψηφία των αγροτών εξαιρούνται τελικά από τις υποχρεώσεις ε, πρασινίσματος. Ε, όσον αφορά τις αγροτικές, ε, τις γεωργικές πρακτικές, αυτές επηρεάστηκαν 13% των αγροκτημάτων που, των εκμεταλλεύσεων που 30% των αγροκτημάτων τα οποία επισκέφθηκε η το ελεγκτικό συνέδριο ακολουθούσαν τις πρακτικές και αυτό το ποστό αυξήθηκε στο 37% οπότε δεν είναι κάτι το αμεληταίο επίσης αναφέρθηκε το ότι μπορούμε να πληρώσουμε για πρακτικές οι οποίες ακολουθούσαν ήδη οι γεωργοί κάτι το οποίο αναφέρθηκε ως ε, πεταμένα λεφτά στην έκθεση ε, όπως είπα όμως δεν επιδοτούμε γεωργικές πρακτικές αλλά την παροχή δημοσίων αγαθών και μέσω υφιστάμενων πρακτικών. Και δεν θα ήταν δυνατόν βεβαίως να τιμωρήσουμε τους αγρότες που ακολουθούσαν ήδη τέτοιες ε, πρακτικές. Οπότε το πρασίνισμα δεν λειτουργεί ως ένα αγροπεριβαλλοντικό μέσο το οποίο αποσμειώνει τους ε, αγρότες ε, και για το κόστος ε, το οποίο έχουν ήδη επομιστεί. Ο γενικότερος στόχος λοιπόν είναι να ανταμείψει την παροχή δημοσίων αγαθών από τις γεωργικές δραστηριότητες και εφόσον ήδη παρέχονται κάποια τέτοια δημόσια αγαθά δεν σημαίνει ότι ζητάμε απαραίτητα αλλαγή κάποιων πρακτικών αλλά βεβαίως θα θέλαμε να μην υπάρξει κάποια επιδίνωση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια βλέπουμε μία γρήγορη αύξηση και εντατικοποίηση της μονοκαλλιέργειας, οπότε πρέπει να σταματήσει νομίζω αυτή η επιδείνωση των πρακτικών. Ε, όπως επίσης τόνισε το ελεγκτικό συνέδριο Κομισιόν ε, συμπέρανε στην έκθεσή της για το 2016 για την πρώτη εφαρμογή του πρασινίσματος πως η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και τους γεωργούς ε, δεν έχει επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση του πρασινίσματος και πολλές από τις αποφάσεις ε, οι οποίες ε, ελήφθησαν ε, για να μεγιστοποιηθεί ακριβώς το περιβαλλοντικό όφελος και βεβαίως προσπαθούμε να απλοποιήσουμε, να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε τις απαιτήσεις του πρασινίσματος και αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα απαγόρευση χρήσης ε, ζυζανιοκτών σε περιοχές οικολογικής ε, εστίασης ε, και βεβαίως αυτό ισχύει αρχές αυτού του έτους και το ίδιο συμπέρασμα είχαμε νομίζω και στην δική μας μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους και είπαμε ότι όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή το πρασίνισμα πριν την εφαρμογή των αλλαγών θα έχει μικρή αλλαγή στις πρακτικές και τους περιβαλλοντικούς στόχους αλλά αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μέσω αλλαγών κάθε υποχρέωσης ειδικά στην μεταρρυθμίση του 2017 που έκανε η Κομισιόν. Τούτων λεχθέντων συμφωνούμε με την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου ότι σε πολλέ χώρε είναι πολύ περίπλοκο το πρασίνισμα και πολύ γραφειοκροτικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο επίπεδο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν ξεκαθάρισε στην ανακοίνωσή τη για το μέλλον τη γεωργίας και των τροφίμων που υιοθετήθηκε το Νοέμβριο πέρσι ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική φιλοδοξία και ότι η τρέχουσα αρχιτεκτονική δεν ταιριάζει με την υψηλότερη φιλοδοξία και Ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η προσέγγισή μας για να αυξηθεί το επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας και άρα μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική που θα βασίζεται στις θετικές εμπειρίες του πρασινίσματος και της πολλαπλής συμμόρφωσης, γιατί εκεί πέρα έχουμε ε, θετικές εμπειρίες και αποτελέσματα και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας θα αποτελέσει τμήμα των μελλοντικών νομοθετικών ε, προτάσεων μας ε, που θα υποβάλουμε γύρω στο καλοκαίρι του 2018 και στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη θα περιγράψουν σε ένα στρατηγικό σχέδιο το πώς θα ακολουθήσουν ακριβώς συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, το νερό, τα εδάφη, την δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και περιλαμβανομένης ακριβώς μιας αίρεσιμότητας ε, των πληρωμών και έτσι θα έχουμε μια εσωτερική λογική που θα περιλαμβάνει και την ε, συνεισφορά στην περιβαλλοντική πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια προσέγγιση για την ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της ΚΑΠ και κοιτάμε ακριβώς πώς θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται περισσότερο στην απόδοση στους ε, διάφορους ε, περιβαλλοντικούς στόχους αντί να συνεχίσουμε την προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα που βασίζεται στην συμμόρφωση με βάση κάποιους κανόνες που έχουν τεθεί με τρόπο ενιαίο στο επίπεδο της Ένωσης. Οπότε ναι, το πρασίνισμα έχει αδυναμίες, έχει και δυνατότητες. Ε, για το μέλλον σκοπεύουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση, να πάμε από την συμμόρφωση στην απόδοση για να ανέβει το επίπεδο φιλοδοξίας της ΚΑΠ στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και ένα σύστημα πιο απλό που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των αγροτών και τις τοπικές ε, περιβαλλοντικές ε, συνθήκες. Αυτά για το μέλλον της ε, ΚΑΠ και το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ωστόσο δεν κατάλαβα από αυτά που είπατε, εάν είπατε ε, τι μπορείτε να αλλάξετε κατά τη διάρκεια αυτή της θητεία, σε αυτή την εντολή, σε επίπεδο ΚΑΠ. και ζηρουργικής πολιτικής. πολιτική. Μέχρι τώρα τους τελευταίους 18 μήνες. Κάνουμε μια σειρά από μελέτες αξιολόγησης και παρακολούθησης για να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα του πρασινίσματος. Και τα όσα σχολιάζει το ηλεκτρικό συνέδριο έχουν, προέρχονται από τις δικές μας τις μελέτες λίγο πολύ. Έχουμε λίγα στοιχεία ωστόσο και πληροφορίες για το πραγματικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του γιατί ιδιαίτερα γιατί ο έδαφος ε, και τα ύδατα θα περάσουν 5-10 χρόνια για να δούμε αποτελέσματα. Συνεχίζουμε αυτή την αξιολόγηση, την παρακολούθηση. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην καλύτερη χρήση των μέτρων που προβλέπει η κατεξουσιδότηση πράξη για την απλούστευση, τη βελτίωση των ε, μέτρων για τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, για την ε, διαφοροποίηση περίοδο 2014-2020 δηλαδή, κυρίως την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση για, τη δυνατό, για τις δυνατότητες και την υποχρέωση του greening. Η Πρόεδρος ευχαριστώ, αλλά αυτό είναι κομμάτι του Omnibus. Δηλαδή από την οικολογική προσέγγιση και το πρασίνισμα δεν βγαίνει τίποτα τελικά ή τόσο πολύ το έχετε απλουστεύσει. Απάντηση. Κοιτάξτε, στον κανονισμό Omnibus έχουν εισαχθεί κάποιες αλλαγές για το πρασίνισμα και τις διατάξεις του. Δύο κυρίες αλλαγέ, καταρχάς μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή της ε, προστασίας της διατήρησης των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων ώστε και στο μέλλον να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το μέτρο σε οργού και να εστιάσουμε στην προστασία των χορτολιβαδικών εκτάσεων για τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις όπως έχουμε προβλέψει από το πρασίνισμα του 2014 Πολλές περιοχές που καλύπτονταν από μόνιμες χορτοδολιβαδικές εκτάσεις περιγράφονται ως μόνιμες και λίγες, πολύ λίγες ρεμπό είναι αρνητικός ο αντίκτυπος σε σχέση με την ποιότητα του εδάφους και την συγκέντρωση ε, άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν η αλλαγή είναι η βελτίωση, με στόχο τη βελτίωση των, της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Επίσης στο Omnibus έχουμε εστίαση στη πρασίνημα, ενεργειακές συγκομιδές, αρρώσιμες, πράσινες εκτάσεις που μπορεί να ενισχυθούν χάρη στο μέτρο αυτό, χωρίς ωστόσο να περιμένω ουσιαστική ανατροπή ως προς τη συλλογική οικολογική περιοχή τη σημαντική αλλαγή ως προς την αποτελεσματικότητα του πρασινίσματος και που σχετίζεται με αυτές τις αλλαγές, όπως ε, σας ανέφερα, ε, προέρχεται κυρίως από την καταξουσιοδότηση πράξη που υιοθετήθηκε πέρσι και εφαρμόζεται φέτος. Η πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ, αλλά θα είστε αύριο στην Γεωργική ή κάποιος άλλος από εσάς. Θα είμαι εγώ παρόν. Καλά, ε, και εμείς βέβαια, και εμείς. Τέλεια, πολύ ωραία. Σούπερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Λαπαγιώβα. Τι σημαίνει για μας. Θα αρχίσω λέγοντας ε, κάτι που είπε και η Κομισιόν, ότι το πρασίνισμα δεν είχε στόχο να αλλάξει πρακτικές καλλιεργητικές, ε, αλλά να βελτιώσει το δημόσιο αγαθό. πιστεύουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βέβαια και ε, το σκέλος της κάπου που αναφέρεται στο κλίμα. Δεν είχαμε άλλους στόχους που πρέπει οπωσδήποτε να ε, επιτευχθούν. Ούτως ή άλλως ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να θέσει στόχους, γι' αυτό λοιπόν οι πρώτες μας συστάσεις αφορούν το γεγονός ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μια συνολική λογική παρέμβαση. Δηλαδή τι θέλει να επιτύχει, ποιοι είναι οι στόχοι και βάσει των στόχων να επιλέξει μέτρα χρηματοδότηση κτλ. που είναι τα πλέον προσήκοντα. Εμείς δεν είχαμε συγκεκριμένους ε, στόχους ε, και είδαμε, διαπιστώσαμε μικρές αλλαγές. Το βλέπετε και στην σελίδα 28. 1,8% διαφοροποίηση όσον αφορά, διαφορά όσον αφορά τη διαφοροποίηση ε, των συγκομιδών πολύ μικρές αλλαγές ε, και όσον αφορά τους ε, ε, πρόσκαιρους και όσον αφορά τους μόνιμους λιμόνες. Επομένως, καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Θέλω να είμαι προσεκτικός βέβαια γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον αλλά εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό θα, αυτό θα συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν, μπορώ να αντισταθώ στο να σχολιάσω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ε, ε, ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την υποχρέωση διατήρησης των μονίμων λιμόνων. Το 2015 και μετά έχουμε σημαντική αύξηση στις ε, προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που έχουμε όσον αφορά τους μόνιμους λιμόνες. Αυτό το περιθώριο του 10% μπορεί να είναι τεχνικό αλλά ε, παρόλα αυτά ε, χρησιμεύει, χρησιμεύσε και έχει μειωθεί στο 5% και στη, στη Βόρεια Ευρώπη. Ε, κυρίως επίσης ε, έχουμε διευρύνει με σημαντικό τρόπο το πεδίο αυτών των μονίμων λιμώνων ώστε να συμπεριληφθούν και περιοχές Natura 2000. Εάν αυτό το 1% το οποίο αναφέρεται σχετίζεται με μία μελέτη που έγινε από ε, κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βασιζόμενη η μελέτη αυτή ε, σε προσωμιώσεις πριν από το 2015 όμως αλλά νομίζω ότι θα πρέπει με προσοχή να παίρνουμε τα στοιχεία αυτά και να μην λησμονούμε ότι εάν και βεβαίως αναγνωρίζουμε την, ε, τον αντίκτυπο στις καλλιεργικές ε, πρακτικές ε, που είναι μικρός, αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά ο μικρός αντίκτυπος οφείλεται και στο ότι πολλοί γεωργοί έχουν τουλάχιστον δύο ή τρεις διαφορετικές σοδιές και καλλιέργειες στην στο, στα χρήματά τους. Νομίζω ότι και ε, αυτό συμβάλλει στο αποτέλεσμα ε, και νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα και εν πάση περιπτώσει καταφέραμε να σπάσουμε τη μονοκαλλιέργεια. Ε, κυρίως σε περιοχές ε, ε, που παράγουν σιτηρά αλλά και άλλα. Θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν εντός του γενικότερου πλαισίου τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Το χειρότερο στην υπόθεση αυτή βέβαια πρέπει να πω είναι ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε εμείς, ούτε οι γεωργοί, γιατί είναι μαζικές επικρίσεις που τυπώνονται κατά του ε, πρασινίσματος. Οπότε τους συναντούμε. Το ελεκτικό συνέδριο. Αξιόλογο το μείγμα λοιπόν. Και τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Κύριε Μπασκού. Το χειρότερο για εσά είναι να έχει χρόνο η Επιτροπή μα. Και τώρα έχουμε χρόνο και πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μην το πάρετε προσωπικά, βέβαια. Ποτέ δεν πρέπει κανεί να το παίρνει προσωπικά. Αλλά σα ρωτώ, εσά που είστε εδώ, τι πρέπει να κάνουμε. Τι μα προτείνετε σε εμά, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Και πραγματι και ειλικρινά περιμένω και ενδιαφέρομαι να ακούσω μια σοβαρή συμβουλή. Τι έχετε να απαντήσετε. Well, it is clear that the level of ambition of greening, when it been introduced... Κοιτάξτε, είναι σαφέ ότι το επίπεδο φιλοδοξία του πρασινίσματο όταν εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβαθμιστεί στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Υπόθηκε αυτό ήδη. Πρέπει να αναγνωριστεί. Ταυτόχρονα και πέραν αυτού, για μας έχει αδυναμίες διαρθρωτικές, είναι περίπλοκο, έχει μια ομοιόμορφη προσέγγιση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι διαφορετικές συνθήκες στα κράτη-μέλη. Και τρίτον, ας είμαστε και ειλικρινείς για τις φιλοδοξίες. Μπορεί να ήταν πολύ ψηλότερο στην πρόταση επιτροπής μεν το επίπεδο των φιλοδοξιών. Υπόθηκε αυτό ήδη. Α, πάντως, περιορίστηκε σημαντικά εντωμεταξύ. Και πρέπει λοιπόν τι φιλοδοξίε αυτέ να τι αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το κλίμα και το περιβάλλον, με πιο απλό τρόπο να δίνουμε λύσει και με μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να έχουμε ένα εργαλείο χάραξη πολιτική αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στι ανάγκε του γεωργού, του περιβάλλοντο σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό προτείνω με την ανακοίνωση του προηγούμενου Νοεμβρίου να αλλάξουμε δηλαδή προσέγγιση, αντί να επιβάλλουμε μια σειρά κανόνων στους γεωργούς, για όλους τους γεωργούς όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωση, να ξεφύγουμε από αυτή την ομοιόμορφη προσέγγιση, να αφήνουμε τα κράτη-μέλη να ορίζουν τον ειδικό του στόχο σε σχέση με τις ανάγκες με τα δεδομένα του περιβάλλοντος και του κλίματος που έχουν το καθένα σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο να επιτευχθεί ο συνολικός ευρωπαϊκός στόχος. Και θα έχουμε μια προσέγγιση όχι βάση κανονών, αλλά βάση αποτελέσματος. Προσαρμόσιμη στις τοπικές ανάγκες. Που πιστεύουμε θα μας επιτρέψει ένα άλμα πρόοδου στην αποτελεσματικότητα και βέβαια στις φιλοδοξίες που θα διατυπώσουμε για το κλίμα. Είναι ευπρόσδεκτη η υποστήριξη της Επιτροπής σας προς την ε, μετάβαση για μια προσέγγιση, σε μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα, τους στόχους. Στόχοι και φιλοδοξίες. Ατμοσφαιρικός αέρας, έδαφος, ύδατα και όχι κανόνες που μπορεί να είναι ένα απαραίτητο βήμα, θυμάμαι που ορισμένοι, ενίσχυσης κλιματικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της ε, κοινή γεωργική πολιτική, αλλά τώρα πια είναι ξεπερασμένο, πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο φιλοδοξιών. Κύριο Τσέλερ. Βλέπω ότι είναι σε μια δύσκολη θέση η Επιτροπή. Το είπε και η Πρόεδρος. Λέμε στα γερμανικά την παροιμία ότι όποιος θέλει να αποξηράνει ένα έλο δεν ε, πρέπει να ρωτάει τα έλη. Ε, λοιπόν τώρα να έχουμε ενώσει στον λόμπι μέσα στην Επιτροπή και να συζητούν. Η καλύτερη πρόταση να ήταν η πρόταση της Επιτροπής δεν θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα. Μια ανίερη συμμαχία μεταξύ των διαφόρων συναδέλφων. στις επιτροπές ε, και βέβαια με τις ε, προσδοκίες στα κράτη-μέλη δεν μπορεί να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε το ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να περάσει το θέμα αυτό προς σε άλλο επίπεδο. Να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους για τα περαιτέρω, γιατί κάποιος τελικά θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη. κακά μαντάτα, αλλά έτσι είναι. Ξεκολουθούμε να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά στο ένα βήμα το πραγματοποιήσαμε. Θα μεριμνήσουμε και στο μέλλον για το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να τρέχουν έτσι τα πράγματα όπως έχουν. Και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει και την διαμόρφωση της μελλοντική κουγουπού μετά το 2020 και κινδυνεύουμε από την επόμενη αποτυχία και το ελεγκτικό συνέδριο δεν θα είναι σε θέση να εξηγήσει πώς καταλήξαμε σε τέτοιο πάταγο με 26 διαφορετικές ενόμες τάξεις. Εν πάση ευχαριστώ. Κύριε Πάσκου. Παλέψατε έντιμα, αλλά αποτελέσματα μετράνα τα ευρήματά μας είναι αυτά πάνω στα οποία θα στηριχθούμε και παρακαλώ και τις ομάδες να κοιτάξουν πώ μπορούμε στο μέλλον να επαναφέρουμε το θέμα αυτό με ακρόαση. Η οικολογική διάσταση είναι κάτι που για το δεύτερο εξάμεινο του έτους το συστήσαμε λίγο και στους συντονιστές. Καλό θα ήταν γιατί δεν έχουμε ανοίξει όλο αυτό το πρόγραμμα για την Ήπεθρο. κύριος Γκερμπράντι το είχε εξαγγείλει, δεν υλοποιήθηκε ωστόσο. Άρα καλό θα ήταν να, το, να φωτιστεί και πάλι το θέμα αυτό. Για να μην χάσουμε την αισθήση μας ένα τόσο σημαντικό θέμα με τόσο κονδύλιο. Κύριος Τσέλερ. Ναι, Πρόεδρε, και νομίζω ότι θα ήταν καλό να συζητήσουμε και το μέλλον του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου και στο, και στο πλαίσιο του η συζήτηση για το μέλλον του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου το θέμα αυτό όσοι δεν ασχολούνται με τη γεωργική πολιτική, ας ε, τους καθησυχάσουμε, δεν αλλάζουν τα ποσά. Λένε οι μεν. Οι άλλοι λένε δεν, ε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, δεν ξέρετε πώς δουλεύει το σύστημα. Όχι, δεν πάει έτσι. Υπάρχει υποχρεωτικό κάπινγκ σε κράτη-μέλη. Υπάρχουν μέτρα ουσιαστικά σταθεροποίησης της αγοράς, υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν φέρνουν κέρδος στην Ευρώπη. Έχουν το τόσο πολύ διωγγωθεί οι εκτάσεις για το κυνήγι, για οτιδήποτε άλλο που έχουν πέσει πάνω οι διάφορες ε, επιχειρήσεις ασφαλιστικές ε, και ούτω καθεξής και έχουν διωγώσει τις τιμές και μετά πάμε σε μονοκαλλιέργεια σε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμως. Κυρία Κάντεμπαχ. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση της ε, Προέδρου να το συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε αυτά μαζί γιατί είχαμε και μία τέτοια έκθεση και βέβαια έχουμε και την έκθεση για τους νέους αγρότες όπου βλέπουμε ότι με τα μέσα που χρησιμοποιούμε ε, ο στόχος να φέρουμε περισσότερους νέους στην Γεωργία ή να αναλάβουν επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνεται και αν θέλουμε να έχουμε και στο μέλλον γεωργία και μικρή ε, κλίμακα στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε ανθρώπου που θα το κάνουν αυτό. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, κάτι το οποίο συχνά λέμε και στους συναδέλφου της Επιτροπής ε, Γεωργίας, πρώτα απ' όλα ο τομέας λέγεται και αγροτική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου και αφορά ακριβώ ολόκληρη την ανάπτυξη της υπαίθρου και οτιδήποτε συνδέεται με αυτό και όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία μοιράζουμε εδώ είναι ένα μέσο κατεύθυνσης, δεν είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα επειδή είμαι αγρότης να λαμβάνω κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνονται εάν πληρούνται κάποια κριτήρια, τηρούνται κάποιοι κανόνες κτλ. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες για να ξέρει ο καθένας το τι πρέπει να κάνει, να καταλαβαίνει αν τα κάνω σωστά λαμβάνω κάποιο πριμ. Αλλά πρέπει να τα εξηγήσουμε δηλαδή ότι επειδή κάποιοι λάμβαναν στο παρελθόν χρήματα δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματο. Γιατί ε, λένε κάποιοι ότι δεν μπορεί να μου υπαγορεύσει εμένα η ε, Ευρώπη. Όχι, να, αυτό ακριβώς ε, κάνουμε. Δηλαδή τα λεφτά ακολουθούν κάποια απόδοση, κάτι το οποίο γίνεται, είναι πληρωμή για κάτι συγκεκριμένο και μετά έρχονται τα ε, λεφτά αφού υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο λέτε πραγματικά είναι τόσο σημαντικό και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ηρωνία αυτή τη στιγμή. Εγώ ευρωβουλευτής και φαντάζομαι περισσότεροι ευρωβουλευτές της Υπέθρου αντιμετωπίζουν το εξή. Έρχονται οι αγρότε και μα ε, ρωτάνε τι θα κάνετε για να μην περικοπεί η ΚΑΠ. Και η ηρωνία είναι ότι στι περισσότερε περιπτώσει οι οργανώσει που έρχονται σε επαφή μαζί μου είναι η αιτία των περικοπών, εάν γίνουν περικοπές, γιατί ακολουθούν πολιτικές που δεν ακολουθούν τις αρχές που ακολουθούμε εδώ μέσα, ότι τα λεφτά πρέπει να πηγαίνουν σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, όχι σε τεράστιες ε, βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις, αλλά έτσι έχει ε, προωθηθεί η πολιτική στην Ιρλανδία τουλάχιστον. Και ε, προς τα εκεί το έχουν σπρώξει οι μεγάλες οργανώσεις των αγροτών και τώρα έρχονται σε μένα και τους άλλους ευρωβουλευτές και λένε πώς, τι θα κάνετε για να μην περικοπεί. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ε, τροπάρι και να ακούσουν το ότι τα λεφτά δεν είναι για μεγάλες εντατικές ε, εκμεταλλεύσεις αλλά για μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που προσθέτουν τη θέμενη αξία στην Ήπεθρο και αναφέρατε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η γεωργία αλλά και η ανάπτυξη της πέθρου. Αυτό πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά. Εγώ δεν θέλω να αφαιρεθούν λεφτά από τον ΚΑΠ, αλλά αν πάνε σε μικρές εκμεταλλεύσεις δεν μένουν στην τσέπη των αγροτών. Τα ξοδεύουν τοπικά, βάφουν τα σπίτια τους, πάνε στον κουρέα. Υπάρχει μια τεράστια δυναμική στην τοπική οικονομία δεν πάει λοιπόν αυτομάτως ε, στους ε, υπόλοιπους ντόπιου, αλλά αν πάει στους σωστούς αγρότες ωφελούνται όλοι οι ντόπιοι και ο πατέρας μου ο οποίος ήταν α, ε, μαραγκός. Αν δεν υπήρχε η Γεωργία θα είχαμε αναγκαστεί να φύγουμε από τη χώρα. Αυτά λοιπόν. Είμαι επιφυλακτικός σε Πολλού ε, τομείς, αλλά όσον αφορά τη γεωργία γίνομαι από ό,τι φαίνεται ευρώφιλος. Η Κομισιόν έχει μία εικόνα ποιο παίρνει τα λεφτά όσον αφορά το πρασίνισμα. Για το πρασίνισμα αυτό, γιατί μεγέθη εκμεταλλεύσεων μιλάμε, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Γιατί το πρασίνισμα εισήχθη χωρίς να αξιθεί ε, το συνολικό ποσό της ε, ΚΑΠ. Έγινε μια εσωτερική ανακατανομή. Οπότε ποιος λαμβάνει τι, ποιο μέγεθος ε, έχουν οι εκμεταλλεύσεις. Έχετε κάποιους αριθμούς. Παρακαλώ. αν κατάλαβα αυτό που με ρωτάτε, αναφέρεστε στις άμεσες πληρωμές ή στις πληρωμές για το πρασίνισμα payments, για το πρασίνισμα. Κοιτάξτε, η εισαγωγή των πληρωμών πρασινίσματος δεν τροποποίησε με ουσιαστικό τρόπο την κατανομή ε, των επιδομάτων στους γεωργούς. Στις ε, 25 τουλάχιστον χώρες ε, 35% ε, των άμεσων πληρωμών εισήχθησαν σε αναλογική βάση ε, επιπροσθέτως του Basic Payment Scheme. και βεβαίως σχετίζονται και με την ε, γη και εν πάση περιπτώσει ε, το θέμα του πρασινισματο δεν άλλαξε καθόλου την κατάσταση για τους γεωργούς όσον αφορά το θέμα αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο τρίτα των αμέσων πληρωμών και δύο τρίτα των πληρωμών ε, πρασινίσματος αφορούν και πηγαίνουν στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις από 50 μέχρι, 100, μέχρι 250 εκτάρια. Αυτή, ε, αυτά είναι τα μεγέθη των οικογενειακών επενδύσεων εκμεταλλεύσεων συγγνώμη, που ε, παίρνουν τις πληρωμές από το ε, greening. Λιγότερο από 5, συγγνώμη, 5 όχι 50, λιγότερο από 5 εκτάρια ε, που είναι 5 με 6% περίπου του συνόλου της γης που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απαντήσω λοιπόν άμεσα στην ερωτήσή σας, η εισαγωγή των άμεσων πληρωμών προσυνδύνατος δεν άλλαξε, δεν τροποποίησε με τρόπο δραματικό ε, ή ουσιαστικό ε, την κατανομή των ε, πόρων. επομένω. η στόχευση εξακολουθεί να είναι στις οικογενειακές εκμεταλλεύσει. Οπότε ε, λέτε ότι αποκρίνονται λίγο πολύ οι πληρωμές του πρασινίσματος με τις ε, άμεσες ε, πληρωμές. Είναι λίγο πολύ το ίδιο στατιστικά. Ναι, ναι. Γιατί για να λάβει κανείς την πράσινη πληρωμή, δηλαδή η πράσινη πληρωμή είναι υποχρεωτικό για όσους λαμβάνουν την βασική πληρωμή και εφόσον συνδέεται στα περισσότερα κράτη-μέλη, ναι, δεν έχει αλλάξει η κατανομή. Σωστά. Μάλιστα. Οπότε τώρα ξέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, την Κομισιόν, τους ε, συναδέλφους. Ε, νομίζω ήταν ε, σημαντικό και θα πρέπει να τα εξηγήσουμε στην πολιτική γεωργία. Λοιπόν, η επόμενη συνεδρία είναι 26 Φεβρουαρίου, η Δευτέρα που έρχεται, λίγη τη συνεδρίαση.